Can Ας ξεκινήσουμε παρακαλώ. Καθίστε αν γίνεται. Καλώς ήλθατε μετά τις ε, θερινές διακοπές. Ελπίζω να περάσετε ωραία τις διακοπές σας. Έχουμε μια συνεδρίαση σήμερα και αύριο όπως ξέρετε με πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αν γίνεται λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, θα ήθελα να σας πω, σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη, ότι λάβαμε από τον εισηγητή του σημείου 6 για την ανταλλαγή απόψεων για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού το αίτημα να φύγει το σημείο αυτό από τη σημερινή ημερήσια διάταξη και να γίνει αυτό αργότερα βάσει του κειμένου εργασίας. Έχουμε χρόνο, οπότε μπορούμε να το κάνουμε. Η αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή Πολιτισμού θα υιοθετήσει τη γνωμοδότησή της τον Ιανουάριο, οπότε έχουμε αρκετό χρόνο πριν ε, συζητήσουμε το θέμα αυτό σήμερα. Αν συμφωνείτε λοιπόν με την πρόταση τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης, θα έλεγα να φύγει το σημείο 6 και με αυτή την αλλαγή να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω κάποιον άλλον κάποιον να θέλει να αμφισβητήσει την αλλαγή αυτή. Πάμε στο σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 20 Ιουλίου. Υπάρχουν τα πρακτικά, είναι διαθέσιμα. Θα ήθελα να σας πω ότι τα πρακτικά θα θεωρηθούν ότι εγκρίθηκαν εφόσον δεν υπάρξουν κάποιες ενστάσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αυτής. Σημείο 3. Έγκριση του σχεδίου χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων της Επιτροπής για το 2010 λάβαμε το σχέδιο χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων της Επιτροπής για το 10 από τη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Προς ενημέρωσή σας το χρονοδιάγραμμα των Επιτροπών ο, ετοιμάζεται από τις ε, υπηρεσίες του Κοινοβουλίου μετά την απόφαση τον της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών και λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παραμέτρων, διαρμηνεί, αίθουσε κλπ. Και βεβαίως και τις δικές μας προτάσεις. Από ό,τι βλέπετε, 11 συνεδριάσεις θα έχουμε. Δευτέρα ή Τρίτη ξεκινούν ή Τετάρτη. Δυόμιση μέρες συνήθως κρατάνε με την εξαίρεση του Φεβρουαρίου που έχουμε μόνο μισή μέρα συνεδρίαση. Το ίδιο και τον Οκτώβριο ε, ε, αλλαγές επίσης έχουμε Οκτώβριο και Νοέμβριο με τρι, τρισήμιση, με τριήμερες συνεδριάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις και άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το σχέδιο έχει εγκριθεί. Προχωρούμε. Σημείο 4. Ανακοινώσεις της Προέδρου. θα ήθελα να σας πω ότι στις 20 Ιουλίου έχει γίνει και μια συνεδρίαση συντονιστών μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι συντονιστές είχαν συμφωνήσει επί μια σειρά προτάσεων που θέλω να σας υποβάλω και που υποβάλλονται τώρα στην Επιτροπή μας προς έγκριση. Πρώτον, σύστημα κατανομής πόντων στις πολιτικές ομάδες και για τις γνωμοδοτήσεις. Οι συντονιστές συμφώνησαν ότι το υφιστάμενο σύστημα κατανομής πόντων που βασίζεται στην μέθοδο DON'T όπως γνωρίζετε θα παραμείνει ως έχει μέχρι ότου συζητηθεί και ενδεχόμενα να θεωρηθεί η μέθοδος αυτή σε μια μελλοντική συνάντηση των συντονιστών. Προτείνουμε, προτείνουμε οι συντονιστές να συνεχιστεί το υφιστάμενο σύστημα και να συζητηθεί αν χρειάζεται στο μέλλον καμία πολιτική ομάδα από τις οποίες ζητήσαμε να, να στείλουν προτάσεις τροποποίησης έστειλε κάποια πρόταση, οπότε δεν υπάρχουν προτάσεις αλλαγή προς το παρόν. Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε και, και προτάθηκε από τους συντονιστές αφορά στην στην κατανομή των εκθέσεων είχαμε μια σειρά εκθέσεων προς εξέταση. Μαδέρα και Αζόρες πρώτον. Την πήρε η Γκουε. Δεύτερη, Ευρωπαϊκή, η πρώτη της Επιτροπής για τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Διαφορετικών Ταμείων ανατέθηκε στους, στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Τρίτη πρόταση τροποποίηση του Περιφερειακού Ταμείου που ανέλαβε, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που ανέλαβε το ΕΛΚ. Κατόπιν γνωμοδοτήσεις. Οι συντονιστές συμφώνησαν να δώσουν τον την γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό του 2010 στην πρόεδρο της Επιτροπής ως συντάκτρια της γνωμοδότησης η γνωμοδότηση για την κινητοποίηση του Ταμείου Λεγής της Ένωσης με την ειδική περίπτωση της Γαλλίας ε, συμφωνήθηκε τότε να αποστελεί μια επιστολή στην Επιτροπή Προϋπολογισμών που εγκρίνει την πρόταση. Το τρίτο θέμα ήταν η γνωμοδότηση του, της αποφάσεως του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού που ανατέθηκε στους πράσινους και συμφωνήσαν επίσης οι συντονιστές να δοθούν τα ονόματα των συντακτών το συντομότερο δυνατό. Το τέταρτο θέμα που συζητήθηκε από τους συντονιστές αφορούσε τα εκκρεμή θέματα από την προηγούμενη, την έκτη θητεία και τις προτεραιότητες για την έβδομη. Οι συντονιστές συμφώνησαν τα εκκρεμή αυτά θέματα να συζητηθούν και να συμφωνηθούν πριν το τέλος του Σεπτεμβρίου. Επίσης, προτάθηκε να εγκριθεί και η επιστολή με τη θέση μας για τα θέματα αυτά μέσα στο Σεπτέμβριο. Επίσης συμφώνησαν ότι αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ακολουθεί το, η γραπτή διαδικασία. Θέλω να σας πω ωστόσο ότι εν τω μεταξύ στις 27 Ιουλίου ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου απίφθινε μία επιστολή σε όλους τους πρόεδρους των Επιτροπών ζητώντας να παράσχουν μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου όλες οι επιτροπές στη διάσκεψη των πρώτων επιτροπών πληροφορίες για τα εκκρεμή ετήσονται με το άρθρο 249 και 66 του κανονισμού. Στην ίδια επιστολή υπήρχε η πρόταση που δεν ήταν υποχρεωτική για τις επιτροπές να χρησιμοποιήσουν οι επιτροπές την διαδικασία screening των εκκρεμουσών εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, τις νέες νομοθετικές προτάσεις και τις επιθυμίες τους για την πρώτη, για την νέα θητεία. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το αίτημα του, πρώτου Κοινοβουλίου, η Γραμματεία προετοίμασε ένα σχέδιο επιστολής που περιλαμβάνει δύο τμήματα. Το πρώτο έχει τα στοιχεία για όλες τις εκκρεμότητες, κάτι που είναι υποχρεωτικό και στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε μέχρι τις 9 Ενάτου. Στην επιστολή αυτή υπάρχει ένα δεύτερο τμήμα που αναφέρεται στα μη υποχρεωτικά θέματα και μπορεί να προσθεθεί αυτό στο πρώτο τμήμα που συμφωνήσαμε στην επιστολή για τον πρόεδρο ή μπορεί να σταλεί αργότερα ανάλογα αν θέλουμε περισσότερη συζήτηση ή να μην σταλεί καθόλου. Να σας πω επίσης ότι το σχέδιο αυτό θα συζητηθεί σήμερα από τους συντονιστές μετά την συνάντησή μας, μετά την συνάντηση της Επιτροπής και θα διανεμηθεί σε όλα τα μέλη αύριο πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Το τελευταίο θέμα που συζητήθηκε και συμφωνήθηκε τον Ιούλιο από τους συντονιστές αφορούσε στην ακρόαση του νέου Επιτρόπου συμφωνήθηκε ε, μια διαδικασία έγκρισης ε, λίγο πιο ελαφριά. Αυτό συμφωνήθηκε και στην διάσκεψη των Προέδρων ε, για τους νέους επιτρόπους. Όπως ξέρετε θα έχουμε μια μισή ώρα ανταλλαγή απόψεων που ελπίζουν να ξεκινήσει στις 4 σήμερα και Πρώτα θα μιλήσουν ε, με τον υποψήφιο οι συντονιστέ και κατόπιν θα γίνει συζήτηση με όλα τα μέλη τη Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια τη συνάντηση των συντονιστών σήμερα θα κάνουμε την αξιολόγηση της διαδικασία αυτή, το οποίο θα συνοψιστεί σε μια επιστολή που θα στείλει η πρόεδρος της Επιτροπής στον πρόεδρο. Αυτά είχαμε συζητήσει με τους συντονιστές τον Ιούλιο. Και εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις από εσά, οι προτάσεις θα θεωρηθούν ότι εγκρίθηκαν από την Επιτροπή μας. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος που έχει επιφυλάξεις, αντιρρήσεις, να συμφωνήσουμε με τις προτάσεις των συντονιστών κατά συνέπεια. Να προχωρήσουμε στο σημείο 5. ψηφοφορίες. Όπως ξέρετε ψηφίζουμε το τμήμα του προϋπολογισμού του 2010 που μας αφορά. Τρίτο τμήμα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τον Ιούλιο συζητήσαμε τη γνωμοδότηση που είχε προτείνει η Γραμματεία, συμφωνήσαμε για τις προθεσμίες για την υποβολή των υπολογιών ε, όταν έληξε η προθεσμία είχαμε λάβει 18 τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Θα τις ψηφίσουμε αμέσως μετά την εισαγωγή, τώρα, σήμερα. Γιατί πρέπει να την ε, υποβάλουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν ψηφίσει αύριο η Επιτροπή. Κάποιες περισσότερες πληροφορίες να σας πω είχαμε μία τροπολογία επί του κειμένου, υπήρχε και μία δεύτερη που αποσύρθηκε, ως συντάκτρια δεσμεύτηκα στην κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα ότι το θέμα που θέτει στην τροπολογία της και που την απέσυρε κατόπιν δεν είναι σύμφωνα με τη φιλοσοφία των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Και ότι το θέμα αυτό θα το εξετάσουμε τους επερχόμενους μήνες της ε, δραστηριότητές μας. Τώρα, οι αλλαγές επί του προϋπολογισμού. Και εδώ όπως ήρθαν δύο τροπολογίες του κυρίου Αλφόνση, ενώ μία τροπολογία του, των κυρίων Μποβέ και Αλφόνση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής. Εσείς ωστόσο θα το κρίνετε αυτό. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία μετά από αυτό. Υπάρχουν κάποια σχόλια? Όχι. Αυτό που ήθελα να πω είναι να προτείνω ε, των χειρών να ψηφίσουμε. Ίσως όμως, κάτι που δεν ελπίζω, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας να χρειαστεί να κάνουμε έναν έλεγχο της καταμέτρησης, οπότε θα χρειαστεί να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Γι' αυτό ο Μιγγέλ μου θύμισε ότι πρέπει να κάνουμε ένα έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων. Yeah, now we are Θα κάνουμε μια δοκιμή. Το λέω αυτό γιατί πολλοί συνάδελφοι είναι και νέοι, όχι μόνο στην Επιτροπή αλλά και στο Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι κάναμε ένα τεστ στο Στρασβούργο, αλλά μπορεί να το ξέχασαν καλοκαίρι ήτανε. Ας το ξαναδοκιμάσουμε λοιπόν. Άρχεται, θα πω, άρχεται η ψηφοφορία, βάλτε την κάρτα σας Ναι, Σα το θυμίζω γιατί στο, στις οδηγίες δεν υπάρχουν σήμα, δεν υπάρχουν... Ε, στο πρώτο αριστερό είναι το ναι. Το δεύτερο είναι το όχι ή το κατά και το τρίτο είναι η αποχή. Τώρα αρχίσαμε να ψηφίζουμε. Αν ψηφίσετε βλέπω λοιπόν πόσοι ψηφίσατε. Πρέπει να βάλετε την κάρτα. Second Yes? Okay. I'm Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Uh, Να το ξαναπώ. Uh, το πρώτο αριστερά κουμπί είναι το υπέρ, το ναι. Uh, το μεσαίο είναι η αποχή και το δεξί είναι το κατά. Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε. Τώρα θα κλείσω. I'm open again. Ξανανοίξω. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. The vote is closed. Εκτός μικροφώνου, πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία Και βλέπετε εκεί τα αποτελέσματα. Άρα είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ευχαριστώ και συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση. Μαθαίνουμε, μαθαίνουμε. Να ψηφίσουμε την πρώτη τροπολογία, τροποποίηση του κειμένου. Τροποποίηση παραγράφου του από την κυρία Τιτσέρα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Έγινε δεκτή. Προχωρούμε. Α, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Και βλέπετε τα πότε. Εγκρίθηκε. Τοπολογίες επί του προϋπολογισμού. Για να το τσεκάρουμε. Μεταξύ των τοπολογιών υπάρχουν δύο που έχουν αποσυρθεί. Η 66-56 του κυρίου Αλφόνση και μία τροπολογία που θεωρούμε ότι δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Όλες οι άλλες τροπολογίες από την 66-59 και που τελειώνει με την 66-58 του μπορεί να την ψηφίσουμε ε, ομού, αν δεν έχετε αντιρρήσει. Αλλά υπάρχουν αντιρρήσει και πηγαίνουμε να ψηφίζουμε μία προς μία. Μόνο το 6658 επ' αυτού θα πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Κωνσταντσα, μήπως μπορείτε να επαναλάβετε αυτό που είπετε. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά για την 6658. Και λέει η πρόεδρος, μπορείτε να ψηφίσουμε για το υπόλοιπο. Όχι, όχι. Θα δούμε τις ε, τροπολογίες μεμονωμένα και ξεκινάμε με την 6659. Υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Πρέπει να ρωτήσω όμως, δεν είναι ποιος είναι κατά και αποχές, δεν πρέπει να ρωτήσω. Τέλος πάντων, εγκρίθηκε. Πάμε στην 6661. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. 6662. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 6663. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6-6-5-6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 66-64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66-69 υπέρ κατά εδώ δεν είμαι σίγουρη. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Ε, δεν είμαστε σίγουροι. Ε, ε ψηφίζουμε για την 66-69 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 29 υπέρ εγκρίνεται. 29 υπέρ, 13 κατά, μία αποχή, άρα εγκρίνεται. 66-56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα Έχουμε την προφορική τροπολογία των πρασίνων. υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρινεται 6668 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66-66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66-67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66-58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν θέλω λοιπόν να πω ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση δική σας όσον αφορά τη 66-60 τροπολογία που από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι αρμοδιότητα της ε, Περιφερειακής Επιτροπής. Κύριος Αλφόνς, Συνεχθήκαμε με τον κύριο Μποβέ για αυτή την ε, τόσο δραματική κατάσταση με τι πυρκαγιέ στον Νότο και είπαμε ότι ανελήφθη αυτή η πρωτοβουλία για βοήθεια εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχουν κάποια επιπλέον μέσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τι χώρε, τι περιφέρειε που έχουν πληγεί για να αντιμετωπίσουν τι πυρκαγιέ. Αλλά αυτό το οποίο δεν είναι τόσο σαφέ είναι το οποίο επιτροπή έχει την αρμοδιότητα, εάν όχι εμεί. Εάν δεν είναι η επιτροπή τη περιφερειακή ανάπτυξη, πού, πού αποσκοπεί αυτή η τροπολογία. Κωνσταντσε Κρέλ. Κοιτάξτε, το ότι θέλουμε να επιδείξουμε αλληλεγγύη και να διαθέσουμε κονδύλια, αυτό είναι διαμφισβήτητο. Μόνο που αυτό γίνεται μέσα από την κανονική διαδικασία από το ε, Ταμείο Αλληλεγγύης και όχι μέσα από τον προπολογισμό. Γι' αυτό λοιπόν επί της ουσίας ε, ισχύει αυτό, αλλά σε λάθος μέρος. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με την Πρόεδρο ότι εδώ δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε και πρέπει όλο να περάσει μέσα από την πεπατημένη του Ταμείου Αλληλεγγύης. Um, uh, Κοιτάξτε, ε, δέχομαι αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και ε, θα ήθελα να δείξω και κατανόηση για τις επιφυλάξεις του κυρίου Αλφόνσης. Εγώ προτείνω να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για αυτή την τροπολογία, έχοντας βέβαια κατά νου ότι αυτή η πρόταση μπορεί να καταψηφιστεί αύριο, αλλά ε, πρόκειται εδώ για μια πολιτική δήλωση που εκφράζει τις επιφυλάξεις που έχουν κάποιοι συνάδελφοι σε σχέση με την κατάσταση που περιγράψατε. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προτείνω να ψηφίσουμε για την 66-60. Κοιτάξτε, θα ήθελα να στηρίξω αυτά που είπε η συνάδελφος η κυρία Κρέλ ότι πρόκειται για μια διαφορετική διαδικασία που αφορά το Ταμείο Λεγγύης και βεβαίως ε, το να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι πρέπει να κάνει για να ε, στηρίξει αυτό το τμήμα της Ευρώπης. Αυτό είναι σωστό και συμφωνούμε, αλλά αυτό δεν εντάσσεται στον προπολογισμό του 2010. Θα πρέπει λοιπόν ε, να το εντάξετε στο Ταμείο Λεγγύης και δεν πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Mm. δεν θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Εγώ, όπως την καταλαβαίνω, την τροπολογία δεν αφορά το Ταμείο Λεγγύης. Είναι ευρύτερη η τροπολογία και ίσως να αφορά περισσότερο την Επιτροπή Γεωργίας περισσότερο από τη δική μας. Ε, δεν είμαι βέβαια κάθετη επ' αυτού. Ε, καλούμε βέβαια να αποφασίσω. Τώρα αν επιμένει ο κύριος Αλφόνσης, ε, ξέρετε όμως υπάρχει και κίνδυνος και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας στο αίτημα που καταθέτετε. Δεν νομίζω ότι είναι σύμφωνο με το πνεύμα αυτή της τροπολογίας το Ταμείο Αλληλεγγύης. Γι' αυτό και σας έλεγα ότι η Επιτροπή Γεωργίας είναι πιο αρμόδια. Αλλά δεν ξέρω είναι τόσο προφανές. Οπότε και εμείς να γνωμοδοτήσουμε καταρχήν και μετά να δούμε τι θα γίνει πλευράς προπολογισμού. Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε, δεν πρέπει να τα μπλέκουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πει κάτι, παρακαλώ, αλλά θα ήθελα ή δυνατόν να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Από ό,τι κατάλαβα, δύο συνάδελφοι ε, είναι, διαφωνούν. Εγώ θα έλεγα να γίνει η δυνατον να κλεισουμε αυτη τη συζητηση απο οτι καταλαβα δυο συναδελφοι ειναι διαφωνουν εγω θα ελεγα να γινει η ψηφοφορια αλλά αυτό που είπε και τώρα ο συνάδελφος ε, χρήσιμο ήταν. Κοιτάξτε, θέλω και εγώ να πω κάτι. Σήμερα συζητήσαμε διαμακρών στην Επιτροπή Προπολογισμών, εγώ είμαι μέλος στην Επιτροπή αυτή, ε, συζητήσαμε για τις, ε, το κοινωνικό ταμείο για τις καταστροφές στην Ιταλία που υπάρχει ένα ταμείο και ο σωστός τρόπος είναι να πάμε μέσα από το Ταμείο Αλληλεγγύης και όχι ε, να γίνουν εδώ τροπολογίες. Κοιτάξτε, οι συνάδελφοι που σχολίασαν από ό,τι κατάλαβα διαφωνούν και νομίζω εκφράζουν και τα αισθήματα πολλών άλλων συναδέλφων. Άρα δηλαδή εντάξει, δεν θα ψηφίσουμε. Δεν θα ψηφίσουμε για την τροπολογία 66-60 γιατί καταλήγουμε ε, στο ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία ε, που θα την κάνουμε ηλεκτρονικά Φόσον τώρα ξέρουμε πώς ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία, είναι η ε, τελική ψηφοφορία των τροπολογιών που συζητήσαμε. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφοφορία. 37 υπέρ, που σημαίνει ότι το πακέτο των τροπολογιών μας εγκρίθηκε. Και κλείσαμε με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμόν 5. Από ό,τι θα θυμάστε, το σημείο υπαριθμόν 6, το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, ε, αποσύρθηκε αυτό, άρα διακόπτουμε για 20 λεπτά. Γιατί είπαμε στον κύριο, στον Επίτροπο Σαμέτσκι, ε, να έρθει στις 4. Διακόπτουμε λοιπόν ε, μέχρι τις 4, αλλά παρακαλώ να ξεκινήσουμε ακριβώς στις 4. Σας ευχαριστώ. Είναι Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να αρχίσουμε τη συνεδρίαση, παρακαλώ καθίστε για να συνεχίσουμε. Όπως ξέρετε, τώρα θα έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με τον υποψήφιο Επίτροπο Παύελ Σαμέτσκι. Θα τον υποδεχθώ, ευχηθώ καλώς όρισε ή στα πολωνικά σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαμέτσκι που ήρθατε στην ε, Επιτροπή Περιφορικής ε, Ανάπτυξης, λέει στα πολωνικά και σύγχυσε στα αγγλικά η κυρία Χούμνα. Υπενθυμίζεται προς όλους ότι επειδή δύο επίτροποι από την τωρινή επιτροπή απεχώρησαν διότι έγιναν ευρωβουλευτές όπως προβλέπεται από την διάσκεψη των προέδρων ε, την απόφαση του Ιουλίου θα έρχονται οι νέοι υποψήφοι επίτροποι να εμφανιστούν και να συζητήσουμε τις επιτροπές. Γι' αυτό και ήρθε στην επιτροπή μας ο κύριος Σαμέτση για να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή απόψεων και όπως προανέφερα θα υπάρξει κάποια αξιολόγηση από τη βάση των ανταλλαγών απόψεων και θα συντάξουμε μια επιτοχή προς ε, την διάσκεψη των Προέδρων η ΔΕ Επιτροπή θα συνταχθεί από τους ε, συντονιστές απόψε. Και τώρα, τη σκητάλη έχει ο υποψήφιος επίτροπο Παύλος Σαμέτσκι για να κάνει μια σύντομη εισήγηση. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου και ευχαρίστησή μου να ανταλλάσσουμε απόψεις γιατί αρμοδιότητα είναι δύο θέματα που πάρα πολύ με ενδιαφέρουν και έχω ασχοληθεί στην σταδιοδρομία μου, δηλαδή την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την οικονομική ανάπτυξη. Έχουν περάσει 20 χρόνια στα οποία έχω ασχοληθεί και από τις θέσεις του Υφυπουργού Οικονομικών πρόσφατα ε, ως μέλος του Συμβουλίου της κρατικής μας τράπεζας. Οπότε θεωρώ ότι έχω τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να μπορέσω να χειριστώ τα θέματα της περιφερειακής πολιτικής. Επίσης, νομίζω ότι έχω την κατάλληλη εμπειρία το ώστε να δώσω μια όθηση σε αυτή την πολιτική για να κάνουμε κάτι, για να ανασχέσουμε αυτή την πορεία της οικονομικής ύφεσης. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι ώρες. Έχουμε την χρηματοοικονομική κρίση και την ύφεση που απέδειξαν πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, πόσο είναι απαραίτητο τον έχουμε, τους θεσμούς, τους πιο αποτελεσματικούς για να μπορούμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη. Αναμένεται να, υπάρχει, να υπάρχουν επιπτώσεις ε, από αυτή την κρίση και αυτό ότι θα χτυπήσει τις κυβερνήσεις και τις περιφερειακές αρχές όσον αφορά ε, αγαθά και υπηρεσίες. Όμως, Έχουμε τώρα και νέε ευκαιρίε, ώστε να κάνουμε τι κατάλληλε διαρθρωτικέ αλλαγέ, να βρούμε νέε πολιτικέ και μέσα, τόσο ώστε να δώσουμε όθεση στην αλλαγή. Και η έκτη έκθεση πρόοδου συνιστά καινοτομία. Θα πρέπει να υπάρχει εξοικονισμό, θα πρέπει να υπάρχει πολυμορφία στην οικονομία, θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή και επομένω είναι παράγοντα σταθερότητα η πολιτική συνοχή. Άρα θα πρέπει με ευελιξία να δούμε τι θα κάνουμε με τι ε, δημόσιε δαπάνε πρέπει να αυξήσουμε, θα πρέπει να αυξηθεί η εσωτερική ζήτηση, η βράχη πρόθεσμη και να έχουμε ταυτόχρονα στόχου επενδυτικού μακροπρόθεσμου. Θα πρέπει να επιταχύνουμε την εφαρμογή αυτών των προτάσεων και να αναλυφθούν κάποιες προσπάθειες, κάποια μέτρα νομοθετικά και μη. Να σας αναφέρω ποιες είναι οι πιο βασικές τέτοιες αλλαγές. Πρώτα-πρώτα, προχρηματοδότηση, προκαταβολή ε, του ύψους των 6,25 δισεκατομμύριων. Δεύτερον, να επιταχύνουμε τις ενδιάμεσες πληρωμές στα βασικά προγράμματα και να διευκολύνουμε τα διάφορα μέσα χρηματοοικονομικής πολιτικής. Τέταρτον, ενεργειακή αποτελεσματικότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά τα σπίτια σε όλα τα κρατημέλη. Επίσης θα πρέπει ξημότητα ε, όσον αφορά τις δαπάνες να γίνει πιο κατανοητή, πιο απλή και να έχουμε ενιαίους συντελεστέ και ε, απλούς συστήματος. Έχουμε την πρωτοβουλία Jeremy θα βοηθήσει τις ε, ΜΜΕ. Οι μικροπιστώσεις επίσης, οι εγγυήσει και τα άλλα μέσα χρηματοοικονομικής πολιτικής. Οπότε το δεύτερο μισό του 2010 θα παρουσιάσουμε μια έκθεση στα πλαίσια του προγράμματος ανάκαμψης. Και γι' αυτό στις 22 Ιουλίου ε, ψηφίστηκε αυτή η πρόταση σαν γενικό κανονισμός. Ζητήσαμε την τροποποίηση του κανονισμού όπου προβλέπονται διάφορα μέτρα για να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράμματος συνοχής. Ε, αυτό θα γίνει με απλούστευση των διατάξεων που διέπουν την πολιτική συνοχή. Σε συνεργασία με τον Επίτροπο Σπίτλα θα συνεργαστούμε και με το Κοινοβούλιο αλλά το Συμβούλιο, τόσο ώστε να εμπληθεί ταχύως η απόφαση για αυτή την πρόταση. Όμως δεν θα χαλάσουμε τις προσπαθειές μας λόγω της απλούστευσης. Όλες οι προτάσεις έχουν περάσει από ελεγκτές, από την Όλαφ, εκπροσώπους του Ελληνικού Συνεδρίου, ούτω ώστε να υπάρχει χρηστή οικονομική διαχείριση. Σας διαβεβαιώνω ότι είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πάρα πολλά ε, λάθη, σφάλματα στην εκτέλεση των προγραμμάτων των διορθωτικών ταμείων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Ο ρυθμός, οι επιδόσεις ε, εκεί υπολείπουν σχέση με τις υπόλοιπες κοινωτικές δαπάνες και γι' αυτό και θα ενισχύσουμε τον εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ρώσο μέλλον της πολιτική Πολιτικής Συνοχής έχει εξελιχθεί στο πρόσφατο παρελθόν για να ανταποκριθεί στις, στη ζήτηση, στις απαιτήσει που υπάρχουν και από την αντιστάθμιση των ε, μείων εκτιμάτων έχουμε φτάσει στο να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τις δυνατότητές μας τους δε τελευταίους μήνες. Έχουμε ένα σωρό συζητήσεις και ευχαριστώ την ε, προκάτοχο διότι έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο. Το 2 Απρίλιο στο Μαριάνσκι Λάζνε οι Υπουργοί Περιφερειακής Πολιτικής σε συνεργασία με μέλη της Επιτροπής σας έκαναν έναν απολογισμό και ε, συζήτησαν για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής και είχαν ως βάση την τέταρτη έκθεση συνοχής του 2007. Κατόπιν είχαμε την ε, έκθεση Μπάρκα του Μαΐου. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να σας τονίζω τα εξή σημεία. Πρώτα πρώτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια επιτροπή από τότε που άρχισε η πολιτική συνοχή, θέλαμε να εξασφαλιστεί ότι η οικονομική ολοκλήρωση θα του καλύψει όλου. Αυτή όμω η ολοκλήρωση που είχε ω όχημα την ενιαία αγορά μπορεί να αποδώσει μόνο εάν όλοι μπορούν να συμβάλλουν και αν όλοι μπορούν να υποφεληθούν. Στα πλαίσια αυτών των προκλήσεων θα χρειαστούμε περισσότερο από ποτέ το να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και των προσώπων αλλά και των περιφερειών. Αυτή η πολιτική βοηθάει στο να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητές μας αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιες συγκεκριμένες και όχι πάρα πολλέ προτεραιότητε, ούτω ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίε και αυτό να το κάνουμε με έναν σφαιρικό, ολοκληρωμένο τρόπο. Η πολιτική συνοχή επίσης έχει συγκεκριμένο τρόπο για να κινητοποιεί όλους τους ε, συντελεστές και παράγοντες σε περιφερειακό το επίπεδο όσον αφορά τις προτεραιότητες. Δεύτερον, χρειάζεται να επικεντρωθούμε περισσότερο όσον αφορά τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Κατόπιν της αξιολόγησης φάνηκε ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν ίσως επικεντρώσει την προσοχή τόσο πολύ όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τη πολιτική. Εγώ θα συνεχίσω το διάλογο με τα κράτη-μέλη, αλλά και τους πανεπιστημιακούς για να διευνήσουμε πώς μπορούμε να ε, αναβαθμίσουμε την ε, επίδοσή μας και να βελτιωθεί η πολιτική μας. Θα προσέξουν περισσότερο τη, τη χάραξη της πολιτικής από τη βάση συγκεκριμένων στοιχείων και θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε προστιθέμενη αξία από την πολιτική μας, αλλά θα προσέξουμε και την εικόνα που δίνουμε προς τα έξω. Τρίτον, χρειάζεται περιφερειακή συνοχή, και υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα μελετήσουμε βαθύτερα και περαιτέρω για να μπορέσουμε να υποφεληθούμε κάποιων επιτευγμάτων όσον αφορά κάποιε τοπικέ αναπτυξιακέ πρωτοβουλίε, προγράμματα όπω το Urban, το Leader, να αυξηθεί ο, η συμβολή των τοπικών περιφερειακών τελεστών, ε, να έχουμε σύστημα διακυβέρνηση με πολλαπλά επίπεδα και να είναι καλύτερη συνεργασία. Αυτές, αυτά είναι τα θέματα τα οποία μας εμπνέων μας προκαλούν και τέλος είναι το θέμα των μηχανισμών της υλοποίηση, γιατί δεν αρκεί να έχουμε αποτελεσματική ε, εκτέλεση της πολιτικής ε, άσκησή της, θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι χρειάζεται νομιμότητα, χρειάζεται κανονικότητα στις ε, δαπάνες. Το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης, το τωρινό και ιδίω. το σύστημα επένδυσης και ελέγχου συμμόρφωση, το σύστημα αυτό το οποίο έχουμε πρόκειται να αποδώσει καρπού στα μέσα επόμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε ακόμη περισσότερο το διοικητικό ε, βάρος, άχθο για τους εκτελεστικούς φορείς αλλά και για τους ε, καλυπτόμενου, του τους από την πολιτική αυτή και αυτό έχει σχέση με τον κοινοτικό προπολογισμό και εδώ πέρα μπαίνει ο ρόλος της νέας συνθήκης της Λισαβόνας ούτως ώστε να μπορέσουμε να περιχαραγώσουμε την πολιτική μας με νομιμότητα και κανονικότητα όσον αφορά τις δαπάνες. Και κυρίω θα πρέπει να αρθεί κάθε αβεβαιότητα στου εκτελεστικού φορεί. Οπότε και χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών, ούτω ώστε οι διατάξει του δικαίου σε κάθε επίπεδο να μπορούν να είναι όσο γίνεται σαφέστερες. Τώρα θέλω να ολοκληρώσω την εισήγηση λέγοντάς σας ποιες είναι οι βασικές μας προτεραιότητες για τους αμέσους επόμενους μήνες. Άμεση πρωτοβουλία, άμεση προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά το ποιες θα πρέπει να είναι οι αλλαγές στο γενικό κανονισμό και αυτό θα ε, θα, θα γίνει με συνεργασία μαζί σα, ε, συνεργάζεται μαζί σα η Γενική Διεύθυνση τη Κομισιόν για την Περιφερειακή Πολιτική, μαζί με την Επιτροπή σα. Θα τα συζητήσουμε. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την αναθεώρηση του προπολογισμού. Οπότε θα έχουμε ένα έγγραφο προσανατολισμού, το οποίο θα σα υποβάλουμε τέλο ε, του φθινοπόρου. θα βασιστούμε στη δουλειά του Φαμπρίτσιο Μπάρκα και του ΟΣΑ και σε άλλα σχετικά έργα και τεκμηρίωση. Τέλος, ε, θα πρέπει να δούμε ότι είναι μεγάλη προτεραιότητα το να συζητήσουμε τα συμπεράσματα των ε, αξιολογήσεων εκ των υστέρων, ex post. Θα έχουμε την πέμπτη ε, έκθεση της συνοχής, καθώς θα έχουμε και την αξιολόγηση που έχει γίνει και έχει ήδη εξεγγίσει αυτή η αξιολόγηση για, για, για το πλαίσιο μέχρι το 2013. Πρώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Θα αρχίσει η συζήτηση και θα δώσουμε πρώτα-πρώτα τους συντονιστές το λόγο, αλλά σας λέω τα εξή πρώτα-πρώτα. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να σα πω ότι ε, με χαρά μας βλέπουμε εδώ ότι είναι ο πρόεδρος Επιτροπής των Περιφερειών, ο κύριος Λίκ Φαν Μπράντε Ευχαριστούμε που ήρθατε να μας δείτε. Και, και επίσης ε, όλους τους ε, ομολόγους μας που προέρχονται από άλλα κοινοβούλια, από άλλες επιτροπές, για να ακούσουν την ανταλλαγή να απόψεων με τον Επίτροπο. προσοχή υπάρχει web stream, δηλαδή μεταδίδεται στο ίντερνετ αυτή η συνάντηση, αυτή η συνεδρίαση, το οποίο σημαίνει ότι όποιος μιλάει τον παίρνει μια κάμερα. Ε, τον φιλμάρει μια κάμερα και τον μεταδίδει, οπότε λάβετε το αυτό υπόψη. Επίσης επαναλαμβάνω ότι υπάρχει αρκετό χρόνος, ούτω ώστε να γίνει μια πλήρης ανταλλαγή απόψεων. Αλλά είναι σαφή τα χρονικά όρια. Οπότε, όταν λάβουν τον λόγο οι συντονιστέ του, παρακαλώ να περιοριστούν ή στο να μιλήσουν. Τέσσερα λεπτά. Ποιος θέλει πρώτος το λόγο. Uh, Ο Γιάννα Ολμπριχτ και μετά η Κωνσταντσέ. Να μιλήσω λίγο στην δική μου και δική σας γλώσσα κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχάς εξ ονόματος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να σας καλωσορίσω και να σας πω ότι με χαρά σας συναντάμε και να ξέρουμε τι θα κάνετε ως μέλος της Επιτροπής. Έχω ακόμα μεγαλύτερη χαρά ως βουλευτής από την παρουσίαση εδώ γιατί είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί σας για πολλά χρόνια και σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα ρωτήσω λοιπόν ποιος είστε, σας ξέρω πολύ καλά. Να σας κάνω όμως μια σειρά ε, παρατηρήσεων ε, στα αγγλικά. Η... Γιατί διευκολύνει την επικοινωνία. Έχω ορισμένε πολιτικού χαρακτήρα ερωτήσει. Πρώτον, κύριε Πίτροπε, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αποτέλεσμα της κρίσης για την πολιτική συνοχή στο μέλλον. Θα δούμε μια ενίσχυση της πολιτικής συνοχής ή θα αποτελέσει, ή θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση των δύσκολων εποχών. Υπάρχει ο κίνδυνος στο μέλλον να, μειώσουμε, να μειωθεί η σημασία της πολιτικής αυτής, ιδίω από τις χώρες που θεωρούνται ως καθαροί πληρωτές. Υπάρχει μια διπλή συνέπεια λοιπόν. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά, διότι αυτό που εσείς και εμείς θα πράξουμε τους επόμενους μήνες θα επηρεάσει το μέλλον. Μια δεύτερη σύντομη ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σας ως προς τον ρόλο του Επιτρόπου σχετικά. Ξέρω ότι απαντήσατε βάσει της συνθήκης. Ποιος είναι ο ρόλος ωστόσο του Επιτρόπου και της Επιτροπής ευρύτερα στην πολιτική αυτή. Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος στην δραστηριότητα αυτή εμπλεκόμενος ο ή επόπτης. Σύμφωνα με και βέβαια και το θέμα που είναι βέβαια τεχνικού χαρακτήρα πώς θέλετε να υπερασπιστείτε την Επιτροπή μπροστά στα επιχειρήματα εκ νέου του ελεκτικού συνεδρίου που θα τονίζει την ανάγκη ε, να έλεγχονται καλύτερα οι δαπάνες, ότι υπάρχουν κονδύλια που δεν αναλύσκονται κτλ. Η παρατήρησή μου είναι ωστόσο η εξή. Στην Επιτροπή τα τελευταία χρόνια είχαμε, στην Επιτροπή μας είχαμε συνεργαστεί πολύ στενά με την Κομισιόν. Πολύ συχνά υπερασπίζαμε τις προτάσεις της Επιτροπής. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Αν είναι δυνατόν και επίσημα. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις του Συμβουλίου για την έκθεση αυτή. Έχουμε τη συζήτηση αύριο, αλλά φαντάζομαι ότι οι προτάσεις σας δεν θα ικανοποιήσουν όλα τα κράτη, δεν θα έχουν ικανοποιήσει όλα τα κράτη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει πρόεδρος, η Κωνσταντσα Κραέλ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ζαμέτσκι, εγώ δεν είχα τη χαρά να σας γνωρίζω παλαιότερα. Γνωρίζω μόνο το βιογραφικό σας, το οποίο είναι εντυπωσιακό πρέπει να πω. Ε, Παρ' όλα αυτά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό το να είναι κανείς επίτροπος ε, για την πολιτική συνοχή από το να εργάζεται σε μια κεντρική τράπεζα. Γι' αυτό λοιπόν επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Είπατε ότι η διαρθρωτική πολιτική είναι σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ε, πράγματι αυτό είναι αλήθεια και εμείς ως Κοινοβούλιο ε, προσπαθούμε να στηρίξουμε κάτι τέτοιο. Μόνο που το θέμα είναι ότι αυτός δεν είναι ο μοναδικός στόχος της πολιτικής συνοχής. Μήπως μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω για τις απόψεις σας για το τι επιθυμείτε να κάνετε κατά τους επόμενους μήνες ε, για την υποστήριξη περιφερειών οι οποίες ε, οικονομικά δεν είναι τόσο προηγμένες. Αναφερθήκατε στην ε, περιφερειακή συνοχή, σε αυτή τη λέξη κλειδί και ρωτώ, επ' αυτού του θέματος προτίθεστε την Άνοιξη να καταθέσετε μία νέα μελέτη και προτίθεστε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θα κάνει η ε, περιφερειακή ή η εδαφική συνοχή. Το Κοινοβούλιο περίμενε η Κομισιόν να καταθέσει μία πρόταση για ορισμό αυτού του όρου ή τουλάχιστον την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί ο όρος. Προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα. Αναφερθήκατε στην έκθεση Μπάρκα και χαίρομαι που ε, θέλετε να αναλάβετε πρωτοβουλίες με βάση αυτήν την έκθεση. Θυμάμαι ότι στην έκθεση αυτή μεταξύ άλλων προβλέπεται μια ομάδα εργασίας η οποία θα προτιμάσει τη μελλοντική πολιτική συνοχής και εκεί γίνεται λόγος ε, για όλους τους θεσμούς που μπορούν να επιτρέπουν, όχι όμως για το Κοινοβούλιο. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε ότι θα υπάρξει μια τέτοια ομάδα εργασίας και επίση ε, φαντάζεστε εσείς ε, σε μια τέτοια ομάδα εργασία να βρίσκονται και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Και έτσι φτάνω στο τελευταίο μου ερώτημα, δηλαδή πώς ακριβώς ε, φαντάζεστε τη συνεργασία με την Επιτροπή. δεν μπορεί να είναι απλά η απόκτηση γνώσεων, θα πρέπει να είναι μια ενεργός συνεργασία. Ε, κατά το παρελθόν το Κοινοβούλιο σας είχε στηρίξει. Εμείς ε, ήμασταν ε, συνεργάτες στη διαμάχη με το Συμβουλίο. Μήπως μπορείτε να φανταστείτε κάτι παρεμφερές για το μέλλον. Αυτές λοιπόν είναι οι πρώτες μου ερωτήσεις και θα ήθελα να μπορούμε να συζητήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι μέχρι το τέλος του έτους. Αλλά ίσως αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε μια άλλη ακρόαση. Για τους ε, φιλελεύθερους, η κυρία Μαλέσκου. Ευχαριστώ, κύριε ε, Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την τοποθέτησή σας στη θέση αυτή. Ακούγοντας την παρουσίασή σας, είμαι πεπισμένη ότι η συνεργασία μεταξύ μας θα είναι εξαιρετικά καρποφόρα και σίγουρα θα βελτιώσουμε την πολιτική περιφερειακή ανάπτυξη τη Ένωση στο εγγύ μέλλον. Η θέση σα σε ό,τι αφορά τι ανάγκε ε, να υπάρχει διάλογο με τα κράτη-μέλη είναι μια σωστή θέση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αρχή της αποτελεσματικότητα στην χρήση των πόρων, αλλά και μια ενοποιημένη συνεκτική πολιτική συνοχή. Θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Πρώτον, η Επιτροπή έχει ήδη τώρα μια σαφή εικόνα για τις περιφέρειες της Ευρώπης που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Υπάρχει μια σαφή εικόνα του ποιε είναι αυτές οι περιοχές και πώς επηρεάστηκαν από την κρίση. Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτηση συμπληρωματικών μέτρων ακριβώς για να βελτιωθεί η δική αυτή κατάσταση και να επιληθούν οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες αυτές. Δεύτερον, τα μέτρα που θέλετε να λάβετε για να προσφέρετε αμέσως ή τουλάχιστον γρήγορα πρόσβαση στα κράτη, στους πόρους για τα κράτη, κράτη που αντιμετώπισαν καταστροφές. Έχετε εξετάσει αυτή τη διάσταση, έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων ώστε τα κράτη αυτά να έχουν μια ευκολότερη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους. Ευχαριστώ και σας Θέλω να σας επιβεβαιώσω εκ νέου τη συνεργασία της ομάδας μαζί σας. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους, ο κύριος Αλφονσί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στη νέα θέση σας και ελπίζουμε η συνεργασία που θα έχουμε μαζί σας στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο γενικότερα να είναι η καλύτερη δυνατή. Δύο ερωτήσεις. Τρεις. Τυπική, επί του τύπου η πρώτη. Το Κοινοβούλιο με, θα έχει εκτεταμένες αρμοδιότητες συναπόφασης και θα χρειαστεί να συνεργαστείτε περισσότερο μαζί μας. Ποια μέθοδο εργασίας θέλετε να υιοθετήσετε. Προβλέπετε έναν κώδικα διοντολογίας. Θα τον υποβάλλετε γραπτός εμείς θεωρούμε ο συντονισμός να είναι εξαιρετικά εκτεταμένος, τόσο ώστε να είναι πλέον επωφελής η ε, από κοινού δυναμικό ανάπτυξης των περιφερειών μας. Επί της ουσίας τώρα η δεύτερη ερώτηση. Είπατε εισαγωγικά ότι πρέπει να απελευθερώσουμε το δυναμικό ανάπτυξη των περιφερειών μας. Διαπιστώνουμε ωστόσο ότι σήμερα λόγω και της κρίσης ανάπτυξη δεν έχουμε. Υπάρχει μείωση της οικονομίας. Εμείς θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανέλθει στην, στο πιστεύω της για την περιφερειακή ανάπτυξη εδώ και δεκαετίες, τη μείωση των ανισοτήτων, την αλληλεγγύη και να αφήσει κατά μέρο τις φιλελεύθερες ε, θέσεις ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Εμείς δεν είμαστε πεπισμένοι ότι η ανάπτυξη αποτελεί απάντηση στην κρίση. Πρέπει να ξαναδούμε την οικονομία, να την ξανασκεφτούμε αν θέλουμε να ε, λύσουμε την κρίση. Το τρίτο ερώτημα αφορά στην θέρμανση του πλανήτη. Ο ΙΕ πριν από λίγο καιρό είχε υιοθετήσει μια έκθεση όπου ανέφερε ότι το 90% των δράσεων κατά του, της ε, υπερθέμανσης του κλίματος θα πρέπει να διεξαχθούν σε υποκρατικό επίπεδο, δηλαδή σε περιφερειακό κυρίως επίπεδο. Η Επιτροπή προτίθεται να προσανατολίσει την περιφερειακή της πολιτική για να λαμβάνει υπόψη καλύτερα την ανάγκη μάχης σε περιφερειακό επίπεδο κατά της υπερθέμανσης του πλανήτη. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους ε, των συντηρητικών, ο κύριος ε, Μπλάσεκ. Πρόεδρε, Χαίρο που μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης. Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου, διότι με τον ίδιο τρόπο βλέπετε το θέμα όπως και εμείς. Προφανώς, για τον τελικό χρήστη πρέπει να απλουστεύσουμε τη διαδικασία, να μειώσουμε το, βι, το διοικητικό άχθος και χρειάζεται ταυτόχρονα να προβλέψουμε τις δυνατότητες ε, λειτουργικών και επιχειρησιακών αλλαγών. Ευελιξία λοιπόν. Το πρώτο ερώτημά μου αφορά αυτό το θέμα. Πρέπει η διαδικασία τροποποιήσεων να είναι όσο απλούστερη γίνεται. Το δεύτερο ερώτημα αφορά τους ελέγχους που γίνονται στην χρήση των πόρων. Η έλεγχη σε κάποια κράτη μπορεί να είναι τεσσάρων βαθμών σε τέσσερα επίπεδα δηλαδή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βάρο. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια απλοποίηση των ελέγχων και εκεί. Τελευταίο ερώτημα. Τα συμπεράσματα που ήδη υποβλήθηκαν στο Μάριεμπαντ. Στο Μαριάν Σκελάζνε. Ναι. Για τις περιφέρειες να εξαντλούν οι περιφέρειες τα τους πόρους όταν δεν, είναι όταν εφόσον ε, έχουν αναλώσει όλους τους πόρους. Και εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει μια φάση phasing out όταν οι, χώρες, οι περιφέρειες δεν έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τους ε, πόρους. Εξ ονόματος ε, της Γκουε, ο κύριος ε, Ελί Ορό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στις ακραία περιφερειακές περιοχές της Ένωσης. Επτά τέτοιες περιφέρειες υπάρχουν. Κανάρια, Αζόρες, Μαδέρα, Γουαδελούπη, Γουιάννη, Μαρτινίκα και Ρενιόν. Με 4 εκατομμύρια κατοίκους σε 25 νήσους με την εξαίρεση της Γουιάννας που βρίσκονται σε όλους τους ωκεανούς της γης. Η ειδικός χαρακτήρα τους σχετίζεται με, τον την ισιωτικότητά τους, την... το γεγονός ότι είναι πολύ μακριά, την ε, ενεργειακή εξάρτηση και άρα η κοινωνική και η οικονομική ευα... τροτότητά τους αναγνωρίζεται από τη συνθήκη μέσω του άρθρου 299 ε, δέλτα τη συνθήκης του Άμστερνταμ. Πέραν αυτών των δυσκολιών ωστόσο, Πρόσφατα κείμενα, πρόσφατες ε, πρωτοβουλίες ε, αποτελούν τροχοπέδι στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών και στην, ε, στον περιορισμό των στόχων που έχουν τεθεί. Φερρυπίν, οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ για τις χώρες της Καραϊβικής υπογράφηκαν οι συμφωνίες αυτές. Σε ό,τι αφορά την μεσημβρινή και Ανατολική Αφρική έχουν συναυθεί την περασμένη εβδομάδα συνάφθηκαν οι σχετικές συμφωνίες. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι είναι απαράδεκτο η διαδικασία αυτή να διεξάγεται και να συνεχίζεται χωρίς την συμμετοχή και την διαβούλευση των περιοχών αυτών της Ένωσης που βρίσκονται στην αντίστοιχη γεωγραφική ζώνη. Θα μπορούσατε κύριε Πίτροπε να αναφέρεται και να υπογραμμίσετε στην αρμόδια για το εμπόριο επίτροπο να εμπλακεί και η υπερπεριφερειακή αυτή δομή στις συναφείς ε, συζητήσεις. Να μιλήσω επίσης και για το διαφοροποιημένο φορολογικό καθεστώς και την ειδική φορολογία που επιβάλλουμε σε προϊόντα που εισέρχονται στην επικρατειά μας και που χρησιμεύουν κυρίως την χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορείτε κύριε Επίτροπε να μας εξασφαλίσετε ότι θα φροντίσετε ώστε να προστατεύσετε για τις περιοχές αυτές το διαφοροποιημένο φορολογικό καθεστώς, ιδίως για τα υπερπόντια εδάφη. Σε ό,τι αφορά την εξάρτηση από τη, τα ορυκτά καύσιμα. Κάποιες από τις περιοχές, ε, από τα νησιά αυτά, έχουν θέσει ως στόχο την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας εντός 25 ετών. Ήδη έχουν ξεκινήσει δράσεις που δείχνουν ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί. Ρωτώ, κύριε Επίτροπε, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι είστε έτοιμος να συμβάλλετε σημαντικά στις περιοχές αυτές ώστε να πετύχουν τους στόχους της οικονομικής απεξάρτησης. Ενεργειακή συγγνώμη απεξάρτησης. Και να τελειώσω, η Σουηδική Προεδρία έχει ένα πλάνο προστασίας και έρευνας της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλασσών και των ωκεανών, ούτως ώστε κάτι τέτοιο να ξεκινήσει γρήγορα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είστε έτοιμος να συνεργαστείτε κύριε Επίτροπε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank ε, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Τζον Μπάφτον. Σας καλωσορίζουμε κύριε Επίτροπε και επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις σχετικά με το πότε θα πρέπει να εκχωρηθούν, να εκταμιευθούν τα κονδύλια στα κράτη-μέλη. Γενικά η όλη διαδικασία είναι πολύ γραφειοκρατική και ε, δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Τα προγράμματα εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο και τα κριτήρια είναι πολύ περιοριστικά. Ε, θα πρέπει όμως να έχετε πάντα κατά νου ότι κατά κύριο λόγο πρόκειται για τα δικά μας χρήματα, τα χρήματα των φορολογουμένων, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Τώρα λοιπόν, εξετάζοντας ε, το ε, κλίμα που επικρατεί και τη χρηματοδότηση εν ώψη της κρίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσετε περιπτώσει όπου δεν θα υπάρχουν χρήματα. Ε, κάποια προγράμματα είναι καλά, αλλά όμως ε, δεν ισχύει αυτά το ίδιο. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να αγωνιστούν για τα κονδύλια. Εγώ θα έλεγα να επανεξετάσετε τα κριτήρια που ισχύουν έτσι ώστε να μπορούν ε, τα κράτη-μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια να επωφελούνται. Αυτό θα είναι πρόβλημα τα επόμενα πέντε χρόνια για πολλά κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό ο κύριος Στογιάννοφ ε, για τους μη εγγεγραμμένους. Και μετά θα ακούσουμε τις ε, απαντήσεις ε, του Επιτρόπου και κατόπιν θέλω να πω ότι αν θέλει κάποιος να μιλήσει να το πει τώρα γιατί ο κατάλογος είναι ήδη μακρύς. Ο κύριος Στογιάνοφ, παρακαλώ. Κανείς δεν θέλει να μιλήσει εξ ονόματος των ε, ανεξαρτήτων. Πολύ ωραία. Ε, να δώσω το λόγο στον κύριο Σαμέτσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ε, με υποστηρίξατε. Σας ευχαριστώ ε, και για την υποστήριξη και για τις ευχές που μου απευθύνατε για το νέο μου αξίωμα. Όσον αφορά τώρα τις ε, ερωτήσεις που ετέθησαν. Η πρώτη ερώτηση θα προσπαθήσω λιγάκι να τις ομαδοποιήσω γιατί είναι δύσκολο να απαντήσω σε κάθε μία ερώτηση ξεχωριστά. Δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα σε σχέση με την κρίση, μια τέτοια ερώτηση, η πολιτική συνοχή σε βράχη πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι επ' αυτού έχω μια σαφή άποψη. Εγώ πιστεύω ότι εν ώψη της ε, κατάστασης όπου η κρίση έλαβε πρωτοφανείς διαστάσεις δεν είχαμε πολλές επιλογές. Ήμασταν αναγκασμένοι να καταφύγουμε στην πολιτική συνοχή ως ένα εργαλείο αντίδρασης. Γιατί αλλιώς οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν πολύ χειρότερες. Γι' αυτό λοιπόν πέρυσι αλλά και φέτος η Κομισιόν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη άρχισε να εφαρμόζει αλλαγές στους ε, κανονισμούς, αλλαγές που θα επιτρέψουν σε μας και στα κράτη-μέλη να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και αποδοτικότητα κατά την εφαρμογή της ε, πολιτικής συνοχής. Ε, γι' αυτό λοιπόν εκπονήθηκαν αυτά τα πακέτα ε, απλούστευσης κατά το παρελθόν. Αρκετά εξ αυτών εξακολουθούν να ισχύουν και ελπίζουμε ότι θα αποφέρουν αποτελέσματα. Βεβαίως τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα ορατά, ε, τα αποτελέσματα καθίστανται ορατά όταν υλοποιούνται τα προγράμματα και όταν αρχίζουν να παρέχονται οι υπηρεσίες και τα αγαθά. Πάντως, οι ρυθμιστικές τροποποιήσεις έχουν ήδη λάβει χώρα. Όσον αφορά τώρα τη δεύτερη ε, πρόταση, η οποία συζητείται πολύ ζωηρά, Δεν μπορώ να πω ότι η πρόταση αυτή ε, στηρίχθηκε ομόφωνα από τα κράτη-μέλη. Όμως, παρόλα αυτά, η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να λύσει κάποια προβλήματα, τα οποία θα αντιμετωπίσουμε κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Από την άλλη βέβαια πλευρά γνωρίζουμε ότι η κρίση ε, είναι στο απογειό της και γνωρίζουμε ότι κατά το δεύτερο εξάμεινο αυτού του έτους και το 2010 ε, αρχίζει σιγά σιγά η ανάκαμψη. Μας περιμένει στη γωνία, λέει χαρακτηριστικά ο Επίτροπος. Δεν μπορούμε λοιπόν να χαράσουμε βράχοι πρόθεσμες πολιτικές, πρέπει να είμαστε πιο οξυδερκείς. Και γι' αυτό, έτσι εγώ θέλω τουλάχιστον, ε, πρέπει να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε το μέλλον της πολιτικής συνοχής και πρέπει να την προσπίστουμε γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλη η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βασίζεται σε κάποιους πυλώνες. Ένας εξ αυτών είναι η πολιτική συνοχής. Αναφέρεται επίσης σε, σε βασικές αξίες της Ευρώπης, ε, στην αλληλεγγύη. Το θέμα όμως είναι πώς όλα αυτά θα λάβουν σάρκα και οστά. Σε αυτή την περίπτωση Θέλω να σας πω το εξής. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτά που ελέγχθησαν από τον κύριο Λαφονσί όσον αφορά τα εργαλεία που πρέπει να ε, εφαρμόζονται, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται. Εμείς την πολιτική συνοχή πρέπει να την χρησιμοποιούμε ως ένα εργαλείο για να εξυγχρονίσουμε ε, τόσο την ευρωπαϊκή οικονομία όσο και αυτή των κρατών μελών και των περιφερειών. Και γιατί, διότι όλο και περισσότερο ε, δεχόμεθα ισχυρή ανταγωνιστική πίεση από άλλα κέντρα σύγχρονης τεχνολογίας, ε, καινοτομιών και αυτό δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν την πολιτική συνοχή πρέπει να τη διαμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι το δικό μας το εργαλείο άμυνας απέναντι στην ανταγωνιστικότητα άλλων περιοχών του κόσμου. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να συνδυάσουμε την αλληλεγγύη με το νέο προφίλ, τη νέα πολιτική η οποία θα πρέπει να ε, στηρίζεται περισσότερο στη συνθήκη της Λισαβόνας από ό,τι μέχρι σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι η στρατηγική της Λισαβόνας εξακολουθεί να ισχύει, δηλαδή εξακολουθούμε να επιδιώκουμε αυτό το στόχο και μετά το 2010 θα πρέπει να αναζητήσουμε μια νέα φάση σε αυτή την ε, πολιτική η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο μέλλον στην πολιτική συνοχής. Και όλα αυτά θα μας ε, βοηθήσουν να αντέξουμε ε, στην πίεση ανταγωνισμού που θα προέρχεται από άλλα μέρη του κόσμου. Υπήρχαν κάποιες ε, πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά την εδαφική συνοχή, γιατί δεν υπάρχει ορισμός μέχρι τώρα για αυτήν. Νομίζω λοιπόν ότι η πράσινη βίβλος σκόπιμα δεν προέβη σε ορισμό της πολιτικής ε, συνοχής. Ζητήσαμε ε, να μας κατατεθούν προτάσεις και από το ευρύ φάσμα απαντήσεων βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση και να πούμε Αντί να προσπαθήσουμε να έχουμε έναν κομψό, ξεκάθαρο ορισμό, να ε, συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που ήδη γνωρίζουμε και που ταιριάζουν μεταξύ τους, όπως παραδείγματος χάρη η συγκέντρωση των ε, πόρων, ε, περισσότεροι πόροι για να προβληθεί η διασύνδεση ανάμεσα στις περιοχές, να υπάρχει μεγαλύτερη συνέχεια και σύνοχη και να υπάρχει καλύτερη διαπεριφερειακή συνεργασία η οποία θα μπορούσε επίσης να προσφέρει και περισσότερες γνώσεις για το πώς ε, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις ε, τοπικές ανάγκες. Νομίζω ότι η συζήτηση από αυτού του θέματος πρέπει να συνεχιστεί ε, και πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση στο μέλλον. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω για άλλη μια φορά αυτό το νέο έγγραφο που σας ανέφερα δεν θα είναι ε, ένα είδος ε, σύνθεσης αλλά θα έχει απλή σύνθεση, αλλά θα έχει ως στόχο να αποτελέσει το σημείο κίνησης για την επόμενη Κομισιόν, η οποία ε, θα πρέπει βεβαίως να χαράξει την πολιτική της από κοινού με το Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα με αυτήν την Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για το μέλλον. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα ε, ποιες ε, περιοχές ε, χτυπήθηκαν σκληρότερα, και κατά πόσο μπορούμε να τους προσφέρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, βεβαίως έχουμε το Ταμείο Λεγγύης το οποίο χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, παραδείγματο χάρη ε, στην περίπτωση του σεισμού του Αμπρούτσο. Προσφέραμε ε, υποστήριξη, το ίδιο μπορεί να γίνει και στο μέλλον. Αν υπάρξουν παρεμφερείς περιπτώσεις που δυστυχώς προκύπτουν. Όσον αφορά τώρα την ε, εδαφική διάχυση επιπτώσεων της κρίσης, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ε, πράγματι εδώ οι γνώσει μας είναι πολύ περιορισμένες. Παρότι υπάρχουν πολύ εξελιγμένες στατιστικές υπηρεσίες που προσφέρουν στην Eurostat και σε άλλους φορείς, παρόλα αυτά πρέπει να βελτιώσουμε τη μέθοδό μας για το πώς ακριβώς εξετάζουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, πώς ε, προσπαθούμε να βρούμε τα μέτρα για να μετρήσουμε την ανάπτυξη και άλλα στοιχεία της συνοχής. Νομίζω ανέφερα ήδη ότι για το μέλλον ένα βασικό στοιχείο είναι η πολιτική συνοχή μετά το 2013. Εγώ είπα ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά ε, το θέμα των ε, exposed ε, αξιολογήσεων, τη μέθοδο, όχι μόνο το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την κατάσταση ορισμένων περιοχών. Πάμε στο θέμα, στο ερώτημα Όσον αφορά το θέμα των ελέγχων και της γραφειοκρατίας που ετέθη το ερώτημα αυτό, εδώ θέλω να σε επισημάνω ένα ζήλημα που υφίσατε. Πράγματι, είναι απαραίτητο, απολύτως απαραίτητο, να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες και οι κανονισμοί που μπορούν να καταστούν ε, απλούστεροι ε, πρέπει να τους καταστήσουμε πράγματι περισσότερο απλούς. Εγώ βέβαια δυστυχώς πιστεύω ότι εξακολουθούμε να έχουμε ένα υψηλό ποσοστό λάθους στις ε, δαπάνες, στους ισολογισμούς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ψάξουμε να βγούμε μια ισορροπία. Βεβαίως και να περιοριστεί η περιττή γραφειοκρατία. Από την άλλη όμως πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν πρέπει με τον τρόπο αυτό να χαλαρώσουν διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε παρενέργειες, δηλαδή λογιστικές ανομαλίες και ακόμα και απάτες. Δεν το έχουμε βρει ακόμα αυτό, το πώς μπορούμε να συμφιλώσουμε με τα δύο πράγματα. Αφενός περιορισμό της γραφειοκρατίας, αφετέρου όμως βελτίωση της, ε, του επίπεδου, της ποιότητας ε, νομιμότητας, οποτεδήποτε εκταμιεύονται κονδύλια ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρόκειται για δημόσιο χρήμα. Όσον αφορά τώρα τις μεταβατικές ρυθμίσεις <coughs> για περιοχές που πάβουν να είναι επιλέξιμες, κοιτάξτε, και πάλι δεν είναι δυνατόν να εισάγει κανείς ε, αλλαγές, όμως ε, στα έγγραφα που προετοιμάστηκαν υπό την αιγίδα, με την βοήθεια της ε, Προέδρου αλλά και σε άλλες εκθέσεις αναφέρονται κάποιοι μηχανισμοί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το είδος των μόνιμων κριτηρίων, αυτά τα μόνιμα κριτήρια πρέπει να εισαχθούν, να είναι ξεκάθαρα, να αφορούν όλες τις περιοχές, γιατί τώρα, πέντε χρόνια μετά τη διεύρυνση, βλέπουμε ότι ε, δεν υπάρχει πλέον ή δεν πρέπει να υπάρχει η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, πρέπει να ισχύουν σε όλες τις περιοχές τα ίδια κριτήρια. Όσον αφορά τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, εδώ πιστεύω ότι η φιλοσοφία της πολιτικής συνοχής ε, τάσεται ανεπιφύλακτα υπέρ αυτών των περιοχών. Δεν πρεπει να υπαρχει ευρωπη των δυο ταχυτητων πρεπει να ισχυουν σε ολες τις περιοχες τα ιδια κριτηρια οσον αφορα τις μόνο για τη συνθήκη, αλλά και για το ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να βοηθάει στην εκμετάλλευση ειδικών χαρακτηριστικών πλεονεκτημάτων. Υπάρχουν βέβαια κάποια ειδικά χαρακτηριστικά ε, που κάνουν δύσκολη τη ζωή αυτών των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών, ακριβώ γιατί είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένε. Υπάρχουν όμω και κάποια ειδικά χαρακτηριστικά όσον αφορά του ε, φυσικού πόρου, το δυναμικό που έχουν για ε, τουρισμό, που είναι σημαντικά. Πρέπει λοιπόν αυτά τα πλονεκτήματα να τα προβάλλει κανείς, έτσι ώστε ε, τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά να ε, διαχέονται σε ολόκληρη την οικονομία μιας χώρας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που δεν απάντησα. Uh, change, uh, uh, Όσον αφορά την ε, κλιματική αλλαγή, εγώ νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή ε, είναι η πρώτη υποψήφια για να γίνει και πρώτη προτεραιότητα στο μέλλον. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία προτεραιότητα όπου θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας αν τελικά συμφωνήσουν όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Νομίζω ότι κάτω από οποιοδήποτε πρίσμα, πολλά έχουν γίνει. Έχουμε πολλά περιβαλλοντικά προγράμματα και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όσον αφορά τα κριτήρια ε, υπάρχουν ε, κάποιες ε, διαδικασίες που οδηγούν στο να αποφεύγονται παρενέργειες, αρνητικές παρενέργειες για το περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι εν μέρη το όλο θέμα έχει αντιμετωπιστεί και όπως σας είπα η κλιματική αλλαγή αδιαμφισβήτητα ε, είναι πρώτη υποψήφια για να γίνει και το επίκεντρο των προσπαθειών μας στο μέλλον. Ένα πράγμα που θέλω να θίξω αφορά στους ελέγχους, γιατί έγινε μια ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία των ελέγχων. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Παραδείγματο χάρη, άκουσα στις συζητήσεις μου με τις υπηρεσίες της Κομισιόν ότι, παραδείγματο χάρη, το ελεγκτικό συνέδριο μερικές φορές εφαρμόζει διαφορετική μέθοδο αξιολόγησης της καταλληλότητας ε, εφαρμογής ε, προγραμμάτων σε σχέση με αυτά που εφαρμόζει η Κομισιόν. Νομίζω λοιπόν ότι είναι φυσικό να μιλάει κανείς, να βρει έναν τρόπο να εναρμονίσει τη μέθοδο με την οποία αξιολογείται η νομιμότητα και η χρησιμότητα ε, των δαπανών. Εδώ λοιπόν υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης σε αυτές τις ενέργειες. Υπάρχει και ένα ερώτημα της κυρίας Κρέλ σχετικά με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μελλοντικές συζητήσεις, σε συζητήσεις για, στο μέλλον για την πολιτική συνοχής. Ε, προφανώς και θα σας ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και θα είμαστε πρόθυμοι να σας ε, καταθέσουμε προτάσεις για να προκαλέσουμε τις ε, συζητήσεις. Στις συναντήσεις ε, μαζί σας, με χαρά μας, θα προσβλέπουμε στις προτάσεις σας προσβλέπουμε στη συνεργασία και στη δική στη συνεισφορά στη συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε τώρα 10 ομιλητές καταγεγραμμένους, οπότε αν θέλουμε να τελειώσουμε όποτε πρέπει, έχουμε το πολύ πολύ τρία λεπτά που μπορεί να μιλήσει ο καθένα, αλλά εάν μιλήσετε δύο λεπτά αυτό θα μας δώσει ένα περιθώριο για παραπάνω ε, παρεμβάσεις. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπή, θα πρέπει να παραδεχθώ ότι με έχει εντυπωσιάσει το βιογραφικό σα αλλά και οι δηλώσει σα. Άρα, θα είστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί τα τέλη του έτου. τέλος πάντων όποια και να είναι, το, το, το, η διάρκεια της εντολή σα. ξέρουμε ότι θα έρθετε στις Βρυξέλλες τώρα σε, σε συγκερούς πάρα πολύ συναρπαστικούς και για σας, αλλά και για την Επιτροπή τη συνοχή. Όπως προαναφέρατε, έχουμε τρία βασικά προβλήματα. Πρώτα πρώτα την οικονομική κρίση. Δεύτερον, έχουμε την όλη προβληματική για την εδαφική συνοχή και επίσης το τι κατεύθυνση θα πάρει η νέα πολιτική συνοχή. Τρίτον, ε, έχουμε κάποιες ε, τελευταίες ειδήσει όσον αφορά τα νέα κριτήρια για την ε, μέτρηση των υπολογισμό των κριτηρίων για τα ευρωπαϊκά ταμεία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το 75% του ΕΠ πρόκειται να μεταβληθεί και θα μεταβληθεί και ο τρόπος καταβολής και εκταμίευσης των ε, πόρων για τις ε, περιφέρειες. Εγώ σας ερωτώ το εξή. Τι φιλοσοφία διαπνέει την πολιτική σας, ποιο είναι το όραμά σας για την ε, νέα πολιτική συνοχή, εδαφική συνοχή σε σχέση με την υπάρχουσα πολιτική. Δεύτερον, ε, τι πρεσβεύεται η δυνατότητα του να μεταβάλουμε τα κριτήρια κατανομής των κονδυλίων μετά το 2013 Νέος προπολογισμός ε, θα γίνει ντόρος, θα γίνει καυγάς μεταξύ των ε, κρατών μελών και άρα εδώ θα διαματεί σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να να συνομιλήσουμε μαζί σα και μαζί να σχεδιάσουμε μια πολιτική συνοχή, η οποία να μπορεί να καλύψει και του 27. Εγώ ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Και τώρα, ερωτήσει εκ μέρου των ε, πολιτικών ομάδων. Σάριος Βόλσκι. Παρακαλώ τώρα, αν μπορείτε. Ε, ε Chairwoman, ε, Τρεις ερωτήσεις έχω κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Γι' αυτό που είπε η συνάδελφος Κρέλ. Είπε ότι είσαστε σαν τραπεζίτης, βλέπω ε, ότι όντως ήσασταν στην Κεντρική Τράπεζα τόσα χρόνια και άλλα 20 χρόνια ήσασταν πανεπιστημιακός. Ασχολούμενος με κάτι σαν την πολιτική συνοχή. Συντονιστή, σε εθνικό επίπεδο και άλλα 10 χρόνια ε, κάθε τη σχετική έρευνα σε πανεθνικό επίπεδο και έχω να σα ρωτήσω μια μπροστά στην άλλη, στην άλλη πλευρά τι συμπέρασματα έχετε αντιλήσει ήσασταν ε, ευεργετούμενος και τώρα θα είστε δωρετής το είπε για την ε, γραφειοκρατία τι είχατε να πείτε για την γραφειοκρατία τη δημιουργία κομισιών Βέβαια και στην επίπεδο υπάρχει γραφειοκρατία και από ό,τι βλέπω ότι είναι 50-50 η ευθύνη. Δηλαδή και η Κομισιόν φταίει αλλά και οι αποδέκτε τη πολιτική. Πολλέ φορέ βέβαια είναι κάτι αναπόφευκτο. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά το να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Για πετε μα, θα πιέσετε τα κράτη-μέλη να σταματήσουν να γκρινιάζουν για την γραφειοκρατία τη Κομισιόν, αλλά να προσπαθήσουν να άρουν και τα, και τα δικά του γραφειοκρατικά εμπόδια. Κάτι το οποίο είναι τόσο βλαπτικό όσον αφορά την ικανότητα απορρόφηση. Τρίτη ερώτηση. Οπότε βλέπω, προσχωρείται στο ρεύμα εκείνο που θέλει η πολιτική της συνοχής να αλλάξει ρότα. Να έχει άλλους στόχους σε σχέση με την πολιτική της συνοχής ε, την οποία οι ιδρυτές της ΙΟΚ εχάραξαν. Μίλησατε για την λυσαγωνοποίηση όπως να πούμε. Τώρα κάπως, κάπως υπερβάλλω, αλλά η ερώτησή μου είναι φοβάστε μπας και απονευρώσετε την κλασική πολιτική που αφορά την συνοχή, δηλαδή την κάλυψη του χαμένου εδάφου. By... Εξίσωση δηλαδή διαφορετικών επίπεδων. Στη στρατηγική της Λισαβόνας, διαχείριση των κρίσεων, ε, μεταβολή κλιματική. Επομένω, τι κάνουμε εδώ πέρα να, να, απομακρυνθούμε από την ε, αρχική φιλοσοφία, απομακρυνόμαστε και από τις συνθήκες και από το πνεύμα των συνθήκων. Κύριε Τρεμόπουλο, έχετε το λόγο. Παρακαλώ προσπαθήστε να τηρήσετε το χρονικό όριο και τον αριθμό των ερωτήσεων όλοι. Ε, κύριε Επιτρόπε, πρόσφατα είχαμε μεγάλες... Πρόσφατα είχαμε μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα που κατέστρεψαν ε, περίπου 20.000 εκτάρια. Για μας υπάρχουν σαφείς κυβερνητικές ευθύνες σε επίπεδο πρόληψης σε επίπεδο δασικής και οικιστικής πολιτικής, μια και ευνοούν τους εμπρισμούς, μη εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών και μη έγκαιρης και αποτελεσματικής καταστολής των πυρκαγιών. Επιπλέον υπάρχουν ακόμη 1.300 ανεξέλεγκτες χωματερές, σκουπιδότεποι, ε, υπάρχει μάλιστα και υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που δημιουργούν μεγάλους κινδύνους και είναι εστίες ε, πυρκαγιών. Επιπλέον, δεν έχουν, ε, αναβάλλονται συνεχώς, ε, δεν ολοκληρώνονται οι δασικοί χάρτες που είναι απαραίτητοι για να διαμορφωθεί και το, να συνταχθεί το, δασικό, το δασολόγιο το οποίο είναι ένα εργαλείο για την υπεράσπιση των δασών και της δημόσιας περιουσίας. Υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του το Σεπτέμβριο του 2007 ζήτησε να επιβεβαιωθεί ότι ε, δεν θα δοθούν οι εκτάσεις που καίγονται για οικοπεδοποίηση ή ε, τουριστικοποίηση και μάλιστα πρόβλεψε να επιστραφούν τα κονδύλια αυτά σε περίπτωση μη εφαρμογής και μη αναδάσωσης ε, των περιοχών. Βεβαίω ρωτώ αν κατά τη γνώμη σας μπορεί να ζητηθεί έλεγχος ε, ή ακόμη και επιστροφή των κονδυλίων σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει ε, αυτούς τους όρους. Να σας πω ότι ε, προτείνουμε να υπάρξει μια αποστολή στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εξετάσει τι ακριβώς συνέβη και τι συμβαίνει. Επίσης, από το Ταμείο Συνοχής θα διατεθούν για την περίοδο 2007-2013 περισσότερα από 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την ε, αντιμετώπιση των ε, κινδύνων των ε, φυσικών καταστροφών. Έχετε υπόψη σας, μπορεί να διαπιστωθεί που έχουν διατηρηθεί αυτοί οι πόροι. Επιπλέον, εσείς με την εικόνα που έχετε, είστε ικανοποιημένος με τον συντονισμό που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών για θέματα προστασίας των δασών, δασοπυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας. Και τέλος, ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόβλημα, ε, πώς θεωρείτε ότι μπορεί να προσφέρει η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόληψη, ε, τι επιπλέον μπορεί, πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια αηφόρα ευρωπαϊκή δασική και οικιστική πολιτική, αν μπορεί να υπάρξει ε, κοινή δράση στην καταστολή των πυρκαγιών, συντονισμός, βοήθεια στην αποκατάσταση μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει και αν το συσχετίζεται όλο αυτό το θέμα των πυρκαγιών, των δασικών με τις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστώ. Έναν ακόμα και μετά θα ζητήσω από το Γιώργο Σαμέτσκι να απαντήσει. Η κυρία Μπριάχ. Συγχαρητήρια κύριε Πίτροπε για, την, για τον διορισμό σας. Με εντυπωσίασαν η παρουσίαση, η παρουσίαση των προτεραιοτήτων που θέλετε να υλοποιήσετε και όπως και εσείς και εγώ εγκρίνω τα μέτρα που υιοθέτησε το καλοκαίρι η ε, κομισιόν για να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση της κρίσης από τις περιφέρειες. Σωστές, ε, σωστά είναι τα μέτρα, αλλά λήφθηκαν κατά εξαίρεση. Άρα είναι προσωρινά εξορισμού. Ωστόσο η αλλαγή των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οικονομικών στοιχείων και δεδομένων θα πρέπει να μας παροτρύνουν να αναθεωρήσουμε βαθύτερα και ήδη από τώρα την περιφερειακή μας πολιτική που συνιστά ένα εργαλείο μίζωνος χαρακτήρα για την οικονομική ανάπτυξη. Εν ώψη της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει κάθε κράτος της Ένωσης, αυτή η αναμόρφωση θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα αντίδραση στην κρίση στην καθημερινότητα. Μήπως ήταν χρήσιμο να υποστηρίξουμε πραγματικά την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιοχών πέραν τη κοινωνική συνοχή και να είμαστε πιο κοντά στην ανάπτυξη και διατήρηση οικονομικών δραστηριότητων επιτόπου. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την εσωτερική τη συνοχή βεβαίω, αλλά να υπερασπίζεται την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια σκηνή για να διαφυλάξει τη βιομηχανία, την οικονομία και την έρευνά μα. Ποιοι είναι λοιπόν οι προσανατολισμοί που εξετάζει η Επιτροπή για να λάβετε υπόψη τις εξελίξεις αυτές στη μελλοντική περιφερειακή μας πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και επίτροπε όσο πιο συνοπτικός γίνεται, αν μπορείτε. Ευχαριστώ. Ορισμός της, περιφερειακής συνοχής, της εδαφικής συνοχής. Όπως είπα, δεν είναι, είναι φευγαλαία η φευγαλαίος ορισμός. Δύσκολα μπορούμε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο. Η δική μου το δικό μου αίσθημα δεν είναι ορισμό, Η δική μου ερμηνεία, αν θέλετε, είναι ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αυτό για να αφαιρέσουμε εμπόδια που προκύπτουν από γεωγραφικές ή από γεωγραφικούς ή εδαφικούς περιορισμούς που αφορούν περιφέρειες, ίσως όχι όλες, όλη την περιφέρεια, αλλά ούτε όλα τα κράτη, αλλά έχουν γεωγραφική αιτιολογία λόγω της τοποθέτησης του, του, που βρίσκονται και με την πολιτική συνοχή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμούς αυτούς. Δεν είναι ορισμός. Η αίσθησή μου είναι όταν με ρωτούν τι άποψη έχω περί αυτού. Όπως είπα, αντί να προσπαθούμε να ε, παρουσιάσουμε μια κομψή προσέγγιση, θα πρέπει να επιδιώκουμε ρεαλιστικές δραστηριότητες που θα ενσωματώνουν την έννοια αυτή της εδαφικής συνοχής στις μελλοντικέ μας δράσεις. Κριτήρια και στοιχεία, κριτήρια επιλεξιμότητας δηλαδή. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον σίγουρα και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι πόροι που θα είναι στη διάθεσή μας θα είναι πάντα λιγότεροι από αυτούς που χρειάζονται. Θα χρειάζεται πάντα να θέσουμε κάποια όρια, κάποια κατόφλια. Αν θα είναι το 75, το 80, το 60 ή το 72,5% εξαρτάται από πολλά πράγματα επιστημονικά στοιχεία, πολιτική διαπραγμάτευση και σίγουρα η νέα επιτροπή θα είναι αυτή που θα εξετάσει πόσο συγκεκριμένα θα πρέπει να αναπτύξουμε και να θεσπίσουμε τις προοπτικές αυτές, τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές ε, μετά το 2013. Ο κ. Σαριουσβόλσκι, ευχαριστώ που διευκρινίσατε κύριε Βόλσκι το βιογραφικό μου. πώς είναι η κατάσταση από την οπτική γωνία των ε, δεκτών της βοήθειας. Πιστεύω ότι δύο μαθήματα μπορούμε να διδαχθούμε. Πρώτον, ο μηχανισμός είναι σύνθετος, όντως πολύ σύνθετος και χρειάζεται απλοποίηση. Δεν μιλώ για την απλοποίηση που αφορά απλούστευση που σχετίζεται με την φυστάμενη κρίση. Αυτή χρειάζεται, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπορούμε να σκεφτούμε έναν ανασχεδιασμό του όλου μηχανισμού που δεν θα είναι τόσο περίπλοκο σαν ένα ελβετικό ρολόι, αλλά θα δουλεύει ταχύτερα, θα παρέχει ταχύτερα αποτελέσματα και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά της νέας επιτροπής των πρώτων ετών της τουλάχιστον. γραφειοκρατία, αν παράγεται από τα κρατημέλη όχι. Κατα... Ε, Προφανώ, εγώ θα καλούσα τα κρατημέλη να μην δημιουργούν γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά δουλειά των κρατών μελών είναι αυτή. Συμβουλέ μπορούμε να δώσουμε. Να του πούμε ότι μην το κάνετε αν είναι περίπλοκο. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στην φιλοσοφία της συνοχής, σχετίστηκε με αυτό που είπε η κυρία Μπριάτ. Με ρωτήσατε, στην ουσία, μήπως πρέπει πρώτα να ξανασκεφτούμε τις διαδικασίες και να κρατήσουμε εσαΐ την απλοποίηση που προσωρινά υιοθετήθηκε. Και το δεύτερο που είπατε είναι η αναθεώρηση της φιλοσοφίας. Και αυτό με φαίνεται σε μια σειρά άλλων ερωτημάτων την πιο σημαντική ίσως ερώτηση. Εγώ δεν απομακρύνω από την αρχική φιλοσοφία. Απλά ο κόσμος εξελίχθηκε, η κατάσταση άλλαξε μετά τη συνθήκη της Ρώμης. Η κατάργηση των υπερβολικών ανισοτήτων δεν σημαίνει μόνο να χτίζουμε δρόμους και να κατασκευάζουμε γέφυρες. Προφανώς χρειάζονται να υπάρχουν κάποιες βασικές υποδομές, δεν τον φυσβητούμε αυτό ιδίως στα νέα κράτη-μέλη, υπάρχουν ακόμα ανάγκες βασικών υποδομών που πρέπει να καλυφθούν. Ωστόσο, αν η Ένωση και στη Δυτική Ευρώπη και στα νέα κράτη-μέλη και στη Βόρεια και στη Νότια Ευρώπη, αν θέλει η Ευρώπη να ανταγωνιστεί με τον υπόλοιπο κόσμο, με τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία, θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε την πολιτική συνοχής και να ενσωματώσουμε σε αυτήν μορφές σκέψης ανάπτυξης των περιφερειών μας που θα τις μετατρέψει σε πιο ανταγωνιστικές. Η βασι, προφανώς η βάση είναι οι βασικές διαθροτικές ανάγκες, αλλά έχουν περάσει έκτοτε 50 χρόνια και πρέπει να σκεφτούμε και την μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε ένα εργαλείο συμπερίληψη στην πολιτική συνοχή για να έχουμε ακριβώ μεγαλύτερη και περισσότερη συνοχή. Για την κατάσταση στην Ελλάδα. Τώρα. Πρέπει να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Την επίγουσα ανάγκη πρώτα. Τα έκτακτα συμβάντα. Υπάρχουν εκεί εργαλεία που μπορεί να μετριάσουν τις πολυτραγικές συνέπειες των δασοπυρκαγιών. Αυτό είναι ξέχωρο. Το ερώτημά σας είναι στην πραγματικότητα κατά πόσο μπορούμε να ζητήσουμε πίσω κονδύλια λόγω της ε, πολιτικής ανεπάρκειας στην Ελλάδα. Δεν είναι δική μας ε, αρμοδιότητα αυτή. Τα κράτη-μέλη, το κράτος μέλος, αν υπάρχει ανεπάρκεια πολιτική σε ένα κράτος μέλος, μόνο την λύπη μας μπορούμε να εκφράσουμε. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Η πολιτική συνοχή παρέχει μια ευκαιρία αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών και να προλαμβάνει στο μέλλον ε, καλύτερα τις καταστροφές αυτές. Αν δεν επιτεύχθη κάτι τέτοιο μέχρι τώρα, αυτό πρέπει να εξετάσουμε από κοινού. Σίγουρα ωστόσο οι ευθύνε δεν είναι στην πλευρά της Επιτροπής και θα καλούσε τις αρχές σας να ξανα να επανεξετάσουν τη στρατηγική και να, να εξετάσουν κατά πόσο αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από Δήμο, από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Επαναλαμβάνω, συναδελφοί. Παρακαλώ, θα βοηθήσει όλο τον κόσμο να είσαστε πιο σύντομοι. Επόμενος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ κύριε Επιτροπέ θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία για τους επόμενους μήνες ή έτη, ανάλογα με το πώς θα προχωρήσουμε. 730 είναι οι ευρωβουλευτές και όλοι πώς να καταλάβουμε τι σημαίνει Δαφική συνοχή. Εμείς εκπροσωπούμε τους λαούς της Ευρώπης που θα πρέπει να μεταλαμπαδεύσουν αυτή την πολιτική στις περιφέρειες και θα πρέπει να δούμε πώς όλη αυτή η υπόθεση, αυτό το όραμα θα είναι μια προσθεμένη αξία για τις περιφέρειες. Ώρες και ώρες τα συζητάμε. Τι σημαίνει τελικά περιφερειακή συνοχή. Εμείς και εμείς το Υπτοκορδιασμοί δεν ξέρουμε. Οπότε πρέπει κάπως να δώσουμε σαν ε, αυτό το όραμα θα πρέπει να το φέρουμε πιο κοντά στον κόσμο, γιατί ο κόσμος περιμένει προτάσεις από την Επιτροπή, προτάσεις κατανοητές. Επίσης, θα σας πω το εξής. Πρώτον, Είπατε, ε, κύριε Επίτροπε, ότι έχουμε σωρό επιδοτήσει που πάνε σε λάθος χέρια και γίνεται λάθος χρήση τους ή κατάχρησή τους. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν πιο απλοί διαγωνισμοί. Γιατί σύμφωνα με έρευνες και μελέτες, ε, όταν δεν εμπλέκονται άμεσα οι περιφέρειες έχουμε τότε περισσότερες λαθροχειρίες. Άρα προσοχή πώς γίνεται η εκταμίευση για να φροντίσουν περισσότερο την υπόθεση που λέγεται περιφερειακή ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε πρώτα-πρώτα βραχυπρόθεσμα τι θα κάνουμε. Κάτι άλλο το που θέλω να σας πω όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια βασικά κριτήρια βασικά κριτήρια αξιολόγηση και να καταλάβουμε περισσότερο και καλύτερα τι θα πει εδαφική συνοχή. Επίσης να έχουμε καλύτερους μηχανισμούς ελέγχου. Να αποκτήσει σάρκα και οστά όλη αυτή η υπόθεση και με ανησυχή η απόπειρα των πράσινων που θέλουν να ε, υπερβάλλουν σε κάποια σημεία ώστε να αποσπάσουν κάποια κονδύλια προσοχή επίσης και στην πολιτική για την ε, αποκατάσταση του κλίματος. Θα πρέπει εκεί να γίνουν επενδύσεις ε, σωστά, να κάνουμε τη διαφορά. Να πάνε τα χρήματα εκεί που υπάρχει περισσότερη βιομηχανία. Επομένως, στο μέλλον, στις προτάσεις της, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ξεχνά ποτέ τον ρόλο της περιφερειακής πολιτικής που έχει σε στόχο και να υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ των διαφορετικών ε, περιφερειών. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Έχει τον λόγο η κυρία Μπέρντε. Έχω μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση. Νομίζω ότι έχει φέρει μια εμπλοκή το Συμβούλιο όσον αφορά την τροποποίηση του Ταμείου Ελεγγύης. Εμείς πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάποια απλούστευση και κινητοποίηση του Ταμείου. Αλλά και διεύρυνση του ρόλου του. Εσείς τι προτείνετε να κάνετε τόσο ώστε να απεμπλακεί αυτή η κατάσταση αδιεξόδου με το Συμβούλιο. Έχω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα για την επικουρικότητα. Ιδίω σε εποχές κρίσης χρειάζονται περισσότερη στήριξη οι Περισσότερη στήριξη από την ΙΟΚ. Άρα να μην ρυθμιστεί αυτό σε εθνικό επίπεδο. Και το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια σύγκρουση με τις εθνικές κυβερνήσεις. Εσείς τι θα κάνετε άμεσα, απευθείας θα βοηθήσετε τις, ε, τις περιφέρειες. Δύσκολο θέμα. Άλλη ερώτηση. Για αυτή την επικάλυψη. Γιατί έχουμε ένα σωρό ταμεία Περιφερειακό Ταμείο ανάπτυξη, αλληλεγγύη, Παγκοσμιοποίησης, Interreg και άλλα και άλλα υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι μερικά από αυτά στοχεύουν να αντιμετωπίσουν κάποιες ad hoc καταστάσεις όπως κάποια κρίση. Όμως, στο μέλλον τι θα κάνουμε, τι θα κάνετε εσείς Επίτροπε, υποψήφιοι Επίτροπε, τρίτη ερώτηση είναι σαφές ότι χρειάζεται απλούστευση. Χρειάζεται να κάτσουμε και να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα χρήματα που πάνε στις περιφέρειες. Σε εθνικό επίπεδο, σε μη εθνικό επίπεδο, γιατί ε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δεν τα πάμε και τόσο καλά και οπότε είμαστε ικανοποιημένοι να έχουμε ε, επίπεδο απορρόφησης 65-66%. Δεν είναι σαφή τα πράγματα. Κύριε Στεξέρα, κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου καταρχήν ε, και εγώ να σας ε, συγχαρώ και να σας ευχηθώ ευόδους των εργασιών σας. Δεν θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Πρόκειται για τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες ε, περιοχές. Γνωρίζω πολύ καλά την ε, κατάσταση στη Μαδέιρα, γιατί προέρχομαι από αυτή την περιοχή. Όμως νομίζω ότι αυτά που ισχύουν στη Μαδέιρα ισχύουν και για τις Κανάριες νήσους. Η Μαδέιρα τα τελευταία 20 χρόνια εξελίχθηκε ιδιαίτερα. Όταν η Πορτογαλία προσεχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Μαδέιρα ήταν στο 40% του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα έχουμε προχωρήσει ε, πολύ πάνω από αυτό. Άρα δηλαδή ε, τα κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν στην Μαδέιρα χρησιμοποιήθηκαν πολύ σωστά. Τα αποτελέσματα των ε, εργασιών τα βλέπουμε και στα στατιστικά δεδομένα που συντάσσονται. Ξαφνικά όμως η περιοχή αυτή υφίσταται σημαντικές περικοπές ε, στα κονδύλια που διατίθενται για την ε, περιοχή αυτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια περιοχή αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξαφνικά όμως η υποστήριξη αυτή συρρυκνώνεται και καταλαβαίνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να συρρυκνωθεί και η ανάπτυξη της περιοχής. Υπάρχει η ε, το άρθρο στη συνθήκη που λέει ότι οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές ε, ε, αντιμετωπίζουν συνεχώ δυσκολίε, άρα δηλαδή ε, χρήζουν και ιδιαίτερη βοήθεια. Θα ήθελα λοιπόν να έχω την άποψή σα κατά πόσον η Κομισιόν είναι πρόθυμη να κάνει μια έκθεση αξιολόγηση, να δούμε κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, οι στόχοι της ε, σύγκλησης ε, έτσι ώστε να ληφθούν και τα απαραίτητα μέτρα στον προπληκτισμό για αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές. Ευχαριστούμε πολύ και κύριε Επίτροπε σας ε, συγχαίρω. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα κάνετε πολύ καλή δουλειά μέχρι το τέλος της νομοθετικής περίοδου. Θέλω να ελπίζω ότι θα παραμείνετε και είμαι σίγουρος ότι τη δουλειά σας θα την κάνετε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά από τη συζήτηση που έλαβε χώρα σήμερα, ε, έχω την εντύπωση ότι η κρίση έσωσε την πολιτική συνοχής. Συμφωνείτε κι εσείς με αυτό. Αν ε, δεν είχε υπάρξει η κρίση, δεν θα υπήρχαν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αλλαγή της ε, πολιτικής. Το τέλος της ε, θητείας της Κομισιόν θα πρέπει να συμπίπτει με την κινητοποίηση όλων των ε, κυβερνήσεων για την βέλτιστη χρήση των κονδυλίων. Παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις και εσείς συμφωνήσατε ότι το μέλλον της πολιτικής συνοχής περιλαμβάνει νέες τεχνολογίες και ε, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα είναι πραγματικά ανταγωνιστικές σε σχέση με την Κίνα, τις Ηνωμένες και τη Βραζιλία. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα μαζί σας, η πολιτική συνοχής πρέπει να στηρίζει την προστασία περιβάλλοντος, όμως ε, αν θέλει κανείς με πολιτική συνοχής ε, να αποκτά περισσότερα κονδύλια θα πρέπει πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα κονδύλια με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και γι' αυτό ερωτώ τις επόμενες εβδομάδες τι προτίθεστε να κάνετε, πώς ακριβώς ε, σκοπεύετε να κινητοποιήσετε τα κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάνει στην Πολωνία η χρήση ε, του Ταμείου των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής, ε, προβλέπεται για τις ε, γέφυρες, τους δρόμους, όλα αυτά που θίξατε κι εσείς. Οι επενδύσεις ε, στην υποδομή δεν λαμβάνουν χώρα όπως θα έπρεπε. Μήπως θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε μια καλύτερη χρήση των κονδυλίων. Η κυρία Μάνερ. αξιότιμο μέλος της Επιτροπής και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ, να σας ευχηθώ τα καλύτερα στη δουλειά που καλείστε να κάνετε. Ε, βέβαια η ερώτησή μου έχει ήδη τεθεί. Θα ήθελα να στρέψετε την προσοχή σας σε περιοχές ε, που βρίσκονται σε μόνιμη μειονεκτική θέση. Υπάρχουν περιοχές ε, που υποφέρουν ε, για γεωγραφικούς, ε, δημογραφικούς λόγους και βεβαίως ε, ένα σημαντικό ερώτημα είναι πόσο μόνιμα θα είναι τα μειονεκτήματα αυτά και πόσο θα λαμβάνονται υπόψη στην πολιτική συνοχή. Πρέπει να συνεχίσουμε να ε, τονίζουμε αυτά τα μειονεκτήματα. Και ποια είναι παρακαλώ η δική σας η άποψη από αυτού κύριε Επίτροπε. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει σχέση με την ε, στρατηγική της ε, Βαλτικής. Αυτό είναι ένα θέμα που ετέθηκα διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας. Πώς μπορεί κανείς να συνδέσει ε, την ε, στρατηγική για τη Βαλτική με την πολιτική συνοχής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείσαμε λοιπόν με τον κατάλογο των ερωτήσεων και θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών να προβεί και αυτός ο κ. Λουκ Βαντεμπράντε σε μία δήλωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχάς να σας συγχάρω για την εκλογή σας. Και το λέω πραγματικά εκ βάθους καρδίας, δεδομένου ότι επιλέξατε να γίνετε μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, σας συγχαίρω και ιδιαίτερα γι' αυτό. Θέλω να πω ότι είμαι πεπισμένος ότι η Επιτροπή σας, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτή η οποία δουλεύει και κάνει ένα δύσκολο έργο να ορίσει πράγματα, ωστόσο τι σημαίνουν στη ζωή ορισμοί όταν δεν υπάρχει πράξη και στην πολιτική, ακριβώς ο στόχος πρέπει εδώ να είναι αν απομακρυνόμαστε ή όχι από τον, το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Προφανώς αλλάζει ο κόσμος και θέλω πρόεδρε να σας ευχαριστήσω εξ της Επιτροπής Περιφερειών. Και λουλούδια, αν θέλετε, μπορούμε να σας δώσουμε για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στην Κομισιόν. Είχαμε μια υποδειγματική συνεργασία ε, μαζί σας τότε και μπορέσαμε να κάνουμε μια σειρά πραγμάτων, όχι, μόσο, όχι μόνο μέσω των επαφών, αλλά και για το μέλλον της περιφερειακής πολιτική. Να σας πω και κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, Είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε τη συνεργασία μας, το ξέρετε, στη ζωή. Καλύτερα είναι να μιλάμε στον κόσμο κατευθείαν και να βρούμε μαζί τους. Αυτό ισχύει και σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών. Κύριε Επίτροπε, καταρχάς να σας συγχαρώ. Σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε τους δεσμούς μεταξύ της Επιτροπής Περιφερειών και της Γενικής Διεύθυνσης. Σίγουρα αυτό μπορεί να γίνει τον Οκτώβριο κατά τη διάρκεια του Open ε, Day, της Open Day. Πιστεύω ωστόσο ότι η εδαφική συνοχή πρέπει να συμπληρώνει τις ελευθερίες των πολιτών και τις ελευθερίες που θεσπίζει η συνθήκη. Προσθέτοντας επιπλέον ε, ελευθερίες, θα υπήρχε το δικαίωμα του πολίτη να επιλέξει που θα ζει και που θα δουλεύει στην Ευρώπη παρά τα εδαφικά μειονεκτήματα. Προφανώς η ελευθερία κυκλοφορίας είναι σημαντική για την Ένωση, αλλά υπάρχει και ελευθερία επιλογής για να αντιμετωπιστούν τα ε, μειονεκτήματα. Κάθε έδαφος πρέπει να στηρίζεται στην αλληλεγγύη της Ένωσης, να μπορεί να στηρίζεται στην αλληλεγγύη της Ένωσης και να προσφέρει στους πολίτες της δυνατότητες καλύτερη ζωή και βελτίωσης της απασχόλησης. Ελπίζω κύριε Επίτροπε να, να συμμερίζεστε το όραμά μας αυτό σε ό,τι αφορά την ε, εδαφική συνοχή και δεν είναι τόσο όραμα όσο προσέγγιση αναζήτηση μιας, ενός τελειορισμού. Τους επόμενους μήνες η Επιτροπή Περιφερειών θα προτείνει στην Επιτροπή να υλοποιήσουμε αυτό το πολυμερές ε, καινοτόμο εργαλείο όπως το αποκαλούμε της εταιρικής σχέσης. Πρόσφατα προτείναμε την προσέγγιση της Λευκής Βίβλου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αυτό το multi-level governance όπως το λένε, και η Επιτροπή και η Κομισιόν ελπίζουμε ότι η Επιτροπή Περιφερειακή Επιτροπή και η Κομισιόν ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουν στο έργο αυτό για να μπορέσουμε στο τέλος του Νοεμβρίου να έχουμε ένα πλήρες κείμενο. Υπάρχει βέβαια και η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού. Τα σύμφωνα εδαφικής συνοχής το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Πρόκειται για τρόπους ενθάρρυνσης μεθόδων διακυβέρνησης που στηρίζονται στην εταιρική σχέση. Ελπίζω κύριε Επίτροπε ότι η Επιτροπή θα συμμερίζεται την αντίληψή μας για τα πράγματα. Τα κοινωνικά ζητήματα θα πρέπει να εμπλουτιστούν χάρη στην ύπαρξη πειραματικών πρακτικών και που θα εκμεταλλεύονται τις γνώσεις και την εμπειρία των εκπροσώπων της περιφέρειας. Αυτό είναι αναγκαίο για να υλοποιηθεί η κοινοτική ε, νομοθεσία σε διάφορες πολιτικές. Και πρέπει να είμαστε σαφείς. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν είναι επαρκώς εμπλεκόμενες στην επεξεργασία των βασικών στόχων που έχουν άμεσες συνέπειες για αυτούς. Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχουμε εμπειρίες, μπορούμε να συμβάλλουμε. Άρα θα είναι αναγκαίο να υπάρχουν νέα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε τη μελλοντική νομοθεσία. Χρειαζόμαστε ισχυρή ε, συνεργασία με την Επιτροπή για να προχωρήσουμε σε καλύτερη διακυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι η κοινοτική περιφερειακή πολιτική θα παράσχει ένα φαινόμενο ταύτισης με την ευρωπαϊκή στρατηγική σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Και ελπίζουμε η Επιτροπή με την συνεισφορά σας, κύριε Σαμέτσκι, να παροτρύνει τη διαδικασία αυτή να, προμο, να προωθήσει την προσέγγιση αυτή και να προτείνει την ανάπτυξη ενός μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης με την Επιτροπή Περιφερειών. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, President. Now the, last uh, point. Uh, Σας ευχαριστούμε. Για τελευταία δέσμη κύριε κυρία Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μέχρι τώρα, από αυτά που άκουσα, είναι σαφές και κυρίω και από αυτά που εσεί είπατε ότι χρειάζεται να κάνουμε το παραπάνω βήμα και να δούμε αν όχι έναν πλήρη ορισμό να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι το οποίο να προσεγγίζει στον ορισμό όσον αφορά την εδαφική συνοχή. Και μπορούμε να συμφωνήσω ότι υπάρχουν κάποιες περιφέρειε που ο κόσμο θέλει μια τέτοια ξεκαθαρή εικόνα. Τι ισχύει, ποιε είναι οι συνέπειε κλπ. Άρα αυτό να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε προς την επίτευξη αυτού του ορισμού. Κάτι άλλο τώρα που αναφέρθηκε. Για την 100% συγχρηματοδότηση είπατε ότι οι περιφέρειες δεν συμμετέχουν οπότε το και δεν ενδιαφέρονται όταν δεν συμμετέχουν για τους διαγωνισμούς θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι κείμενες διατάξεις τηρούνται ακόμα και όταν δεν ισχύει μια τέτοια συγχρηματοδότηση. Θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, όπως γίνεται και τώρα. Για όλους. Πολλές φορές είναι βέβαια πολύ τα πράγματα, πρέπει να τα απλουστεύσουμε. Αλλά θα πρέπει η νομοθεσία να τηρείται. Τι άλλο να πω. Για την αλλαγή του κλίματος, όπως πρόκειψε και από αυτή την ερώτηση, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικοί στόχοι. Τρώσουμε φορά το Ταμείο Ελεγγύης, τα του Συμβουλίου, Είδατε τι έγινε ζητήσαμε να υπάρξει μια φρέσκια πρόταση ε, σε συνέχεια το όσο διαμορφώθηκε το 2005 κάτι να γίνει ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί και η πορεία της γρήπης Ιτανιανίανα τώρα για, τις, ε, για την ε, απότερη περιφέρεια και τα σχετικά επαναλαμβάνω αυτά τα οποία σας είπα. Η Επιτροπή της Συνοχής θα πρέπει να στηρίζεται στα συγκεκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν κάποιες περιφέρειες υπό διαφορετικές μορφές. Είτε είναι φυσική πόρη, είτε είναι γεωγραφική θέση, αλλά υπάρχουν τέτοια συγκεκριτικά πλεονεκτήματα και αυτή είναι η δουλειά της πολιτικής αυτής του, του Δηλαδή πώς θα βοηθήσει τις ε, ε, περιφέρειες, πώς θα τους δώσει δυνατότητα να αναπτύξουν τι οικονομικέ δραστηριότητε. Και έτσι να μεγιστοποιείται το όφελο του κόσμου. Τώρα όσον αφορά την σύγκληση το στόχο 1 του χρόνου θα έχουμε την πέμπτη έκθεση της συνοχής οπότε και θα έχουμε και μια πλήρη αξιολόγηση για τις δραστηριότητες και για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας μέχρι τώρα. Έχουμε άλλε τρεις ερωτήσει του κύριο Μπέρντεν για τις αντιφάσεις, ε, τη σύγκρουση περιφερειών, κρατών μελών και πώ αυτά θα συμβιβαστούν, θα συμφιλειωθούν. Αυτό είναι θέμα κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν. Δεν μπορούμε εμεί να επιβάλλουμε τι προτεραιότητε. Θα πρέπει να το κάνουν αυτό τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ποιο βαθμό τηρούν τι προτεραιότητε των περιφερειών, αυτό τι να σα πω. Τώρα για την επικάλυψη των διαφορετικών ταμείων δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό το σημείο μαζί σας. Θεωρώ ότι οι στόχοι είναι διαφορετικοί του κάθε ταμείου από το άλλο. Το Ταμείο Κοψιμοποίησης έχει δουλειά να βοηθήσει κάποιες ε, περιφέρειες να αντιμετωπίσουν συνέπειες της ε, παγκοσμιοποίηση. Τι αρνητικέ δηλαδή ουσιαστικά την αύξηση τη ανεργία. Αλλά α πούμε το Ταμείο Ελεγγύη είναι κάτι διαφορετικό. Α, όπω είπατε για το Αμπρούτσο, για τι δασοπυρκαγιέ, σε τέτοιε περιπτώσει το επικαλούμαστε. Στα πολωνικά. Σας καλά ε, σας λόγια και για το πόσο βόθησε το Ταμείο όσον αφορά την ε, κρίση. Βεβαίω και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια απλούστευση Και η απλούστευση θα πρέπει να έχει έναν ορίζοντα παραπέρα από την εντοπίση της κρίσης. Αλλιώς έχει επιδράσει η κρίση σε κάθε χώρα. Σας είπα ότι έχω εμπειρία σε αυτά τα θέματα στα αγγλικά τώρα. Βαλτικές χώρες. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το πράγμα που φέρατε. Το πώς λέτε θα εφαρμόζονται οι αρχές της συνοχής σε μια μικρή ομάδα χωρών, υπερφεριών και έτσι να δούμε πώς μπορούμε να ασκήσουμε την πολιτική μας ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάποια σαφής, ε, ε, σαφής ορισμός. Η στατική για την Βαλτική είναι ένα εγχείρημα το οποίο έδειξε και απέδειξε ότι είναι δυνατόν να έχουμε ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων με κάποιον μακρόπνο ορίζοντα, με κάποιον μακρόπνο στόχο. Οπότε, να έχουμε συντονισμό διαφορετικών τομεακών πολιτικών, στήριξη από τον κοινωτικό προπολογισμό και έτσι φαίνεται ότι οι εθνικέ κυβερνήσεις δυνατόν να βοηθήσουν σε διαφορετικά επίπεδα τόσο ώστε να έχουμε ένα, μια άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων. Θα το δούμε τους καρπούς αυτές τι προσπάθειε τα μέσα επόμενα χρόνια. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Επιτροπής, τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών. Νομίζω ότι συμμεριζόμαστε τους στόχους, πολλά πράγματα και άλλωστε ο πρόεδρος Μπαρόσο σας απάντησε ε, με την επιστολή όσον αφορά την λευκή βίβλο για την ε, διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγάλη προσοχή παρακολουθεί αυτή την προβληματική, τις ε, διαβουλεύσεις που γίνονται. Δυναμικά, επομένως, συμμετέχουμε σε αυτή την προβληματική και εντείνουμε τις προσπάθειές μας και τις δραστηριότητές μας. Τέλος, να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα που με βοήθησε πάρα πολύ, με διαφώτισε. Είδα ότι υπάρχουν διάφορες διαφορετικές ιδέες που δεν είχα υπόψη μου. Να είστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα λάβω υπόψη. Εννοείται ότι Όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας και ως Επιτροπή και ως ε, βουλευτές ατομικά. Τα οποία ισχύει βέβαια και για την Επιτροπή των Περιφερειών και σας ευχαριστώ για τη σημερινή συνάντηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ θερμά τον υποψήφιο Επίτροπο για τον χρόνο μα διέθεσε για αυτήν την τόσο παραγωγική συζήτηση και επίση θέλω για άλλη μια φορά συνάδελφοι να σα πω αλλά και να πω και στον υποψήφιο τρόπο ότι τώρα έχουμε συνάντηση των συντονιστών οπότε θα γίνει και η αξιολόγηση τη τωρινή συζήτηση, τα δύο αποτελέσματα πρόκειται να σα υποβληθούν ε, υπό τη μορφή μια ε, επιστολής προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και η ψηφοφορία για την έγκριση της, του ορισμού του κ. Σαμίτσικη ως ε, επιτρόπου θα γίνει στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Πέρα τη συνεδρίαση συνεχίζουμε σε 9 η ώρα αύριο εδώ στην ίδια αίθουσα ώστε να συνεχίσουμε τα θέματα τη επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξη.